Καλησπέρα, 7 λεπτά καθυστέρηση. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Λοιπόν, έκθεση στρατηγική τη ενιαία αγορά. Λάρα Κόμι, εισηγητρία. Δίνω το λόγο στην εισηγητρία. Μετά στου Κιώδη και μετά στου υπολείπου. Χαιρετίζω 20 νέους φοιτητές που έχουν το Κροατία, Πολωνία, Σλοβακία και Ιταλία και είναι εδώ, στην αίθουσα. Καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε. Και 15 νέους έχουμε στα ΖΙΕΡ της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης που είναι εδώ στην αίθουσα. Γεια σας. Η Λάρα Κόμη έχει το λόγο, η Ευχαριστώ Πρόεδρε θα μπορέσουν να ακούσουν οι φοιτητέ και τα πράγματα που είναι ε, ε, τη στρατηγική τη ενιαία αγορά. που να χρησιμοποιήσουν. Και θα ξέρουν από πριν τι θα γράψουν οι εφημερίδε επόμενε μέρε. Έγινε έξοχη δουλειά. Παρουσιάστηκαν πολλέ συμβιβαστικέ. 23. Άρα, συνεπάγεται κατηστρόφω, υπάρχει συνεργασία σε πολλά σημεία. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά και τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει, όσον αφορά την ανάπτυξη της Ευρώπης και την άρση των φραγμών και των εμποδίων που έχουν εντοπιστεί. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες για τις συμβαστικές. Όλοι έχετε το κείμενο. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Όσον αφορά βασικό σημείο άλλο, συμφωνήσαμε τελικά. Με το ECR για το ΦΠΑ. Είναι βασικό σημείο. Key point. Βρήκαμε συμβιβαστική λύση. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Στηρίξαμε και σειρά διαδικασιών προς απλούστευση όλων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μικρομέσες επιχειρήσεις πέρα από την προστασία των καταναλωτών με ένδειξη προέλευσης των προϊόντων. Made in με άλλα λόγια. Και μια άλλη πτυχή που είναι σημαντική για μας να διευρύνουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Κάτι άλλο λειτουργικό, θέλαμε να βρούμε κοινού ορισμούς, ούτω ώστε να ξέρουμε τι είναι νεοφυής επιχείρηση, startup, τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση, πώς μπορούν να εντοπιστούν οι, διάφοροι συμμετέχοντες. Λοιπόν, πάμε και στο sharing economy, στην, στην κοινή οικονομία και στην ψηφιακή ενίαγορά, και επιτευχθέντες συμβιβασμοί νομίζω οδηγούν στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και η ψηφορία θα λάβει χώρα αύριο. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν συζήτηση μαζί με τους άλλους κοιόδης. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Υπήρξε πράγματι πολύ λακωνική. θα δώσω το λόγο στους κοιόδης ξεκινώντας από την μαλεμίτση του S&D. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λάρα και τους άλλους και ηγητές για την συνεργασία τους και τον συντονισμό που είχαμε για αυτή την στρατηγική σημασία έκθεση. Εγκάρδια η ατμόσφαιρα και βέβαια είχαμε πολλές πολιτικές ομάδες που είχαμε διαφορετικούς στόχους αλλά όλα καλύφθηκαν από αυτήν την έκθεση που είναι υποφελής για όλες τις πολιτικές ομάδες αλλά υποφελής και για την έννοια αγορά. Και Έχουμε τις συμβαστικές ως δέσμη. Μας καλύπτουν όλους, φυσικά όχι 100% μιλώντας από πλευρά σοσιαλδημοκρατών. Ε, νομίζω ότι πετύχαμε ένα πολύ ισορροπημένο αποτέλεσμα. Και αυτό πιστεύω ότι θα αποδειχθεί στην ψηφοφορία. Είχαμε λίγο χρόνο, σφιχτόμουν διάγραμμα, δεν συζητήσαμε όσο θέλαμε να τα συζητήσουμε, αλλά προσαρμοστήκαμε, τα έχουμε συνηθίσει. Επίσης, παρά το ότι πολλές μας τροπολογίες καλύφθηκαν από τους αξιόλους συμβασμούς, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και κάποια σημαντικά ζητήματα για τους ε, σοσιαλιστές που δεν πήγαν εκεί, δηλαδή Ρίφιτ, καλύτερο κανονισμό, το διαβατήριο, λιανική, κοινωνική οικονομία, τα οποία δεν καλύφθηκαν. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το πνεύμα στο οποίο κινηθήκαμε, καταλήξαμε σε αυτό το σούρμενο αποτέλεσμα που το βλέπετε στις συμβαστικές και αύριο θα γίνει η ψηφοφορία για αυτήν την ισορροπημένη σταθμισμένη έκθεση. Ευχαριστώ. πρώτος και το λόγο έχει ο κύριος Ντάλτον που είναι ο σχεδόν για την ECR. Και εγώ πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί δούλεψε πολύ και είχαμε πολύ εργαστή συνεργασία οι πολιτικές ομάδες. Από πλευρά ECR θα εγκρίνουμε το τελικό κείμενο, ούτε εμείς πετύχαμε 100% όσα θέλαμε, αλλά είναι καλή συμβασμή και αγκαλιάζουν τις θέσεις μας σημαντικά. Από δική μας πλευράς υπάρχουν κάποια σχετικά για την καινούργια μορφή οικονομία, sharing economy και θεωρούμε ότι τώρα θα υπάρχει ευελιξία οπότε καταναλωτές και εργαζόμενοι θα καλυφθούν και θα προσαρμοστούν στους ρυθμούς ανάπτυξης του 21ου αιώνα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα, να δούμε ε, ε, τι θα γίνει με τον κανονισμό. Πάντως η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ε, είναι το κλειδί για το μέλλον. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι πάντως ακριβώς αυτό, ότι ωφελεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρές η ενιαία αγορά. Έχουν οικονομίες κλίμακας μεγάλε επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Άρα ε, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η προκατάληψη ότι η ενιαία αγορά τι μεγάλες επιχειρήσεις ευνοεί. Άρα θα πρέπει να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που να ωφελεί και τους μικρότερους. Οπότε είναι θετικέ αυτέ οι συμφωνίες και εγώ συμφωνώ ότι για τον ΦΠΑ είναι πολύ σημαντική συμφωνία και επίσης αγωνίστηκε το δικαίωμα στα κρατημέλη να επιβάλλουν να εισπράττουν τον ΦΠΑ τα ίδια, άρα και εδώ πράσινο φω. Υπάρχουν τώρα κάποια που δεν μπορούμε να τα εγκρίνουμε ω πολιτική ομάδα. Βέβαια, το σύνολο τη έκθεση, ναι, θα το εγκρίνουμε. Απλώ εκεί που λέει για την ε, εποπτεία τη ασφάλεια των προϊόντων, ε, εδώ πέρα υπάρχει μια δέσμη διατάξεων που μας βρίσκει μόνος αλλά η υποχρεωτική ένδειξη χώρας προέλευσης δεν μας αρέσει. Πολλά προϊόντα έχουν ε, συστατικά από περισσότερες χώρες. Άρα αυτό ούτε προσθέτει τον καταναλωτή και θα είναι και δύσκολο, ούτε θα είναι ανιχνεύσιμο, ούτε θα ωφελήσει όσον αφορά τις απομιμήσεις και παραποίησεις. Ε, άρα δεν θεωρούμε ότι η υποχρεωτική ε, επισήμανση πρόκειται να κάνει κανένα καλό στην αγορά. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα σήματα που έχουν προπλασιαστεί. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από την κατάτμιση, τη σύγκριση του καταναλωτή, τι επιχειρήσει από παραπάνω δαπάνε. Ε, αυτά για την επισήμανση τώρα. Ε, um, uh, Τώρα για τα προϊόντα που δεν είναι γεωργικού χαρακτήρα θα πρέπει να δούμε εάν θα καλυφθούν. Γιατί αυτά τα προϊόντα, όταν είναι γεωργικού χαρακτήρα, καλύπτονται από τους οργανώσεις των παραγωγών. Όμως όταν δεν είναι, αυτές οι γεωγραφικές ενδείξεις, ναι. όταν αφορούν τη γεωργία, καλύπτονται από τις, από τις πλατφόρμες της γεωργίας. Αλλά θα πρέπει να δούμε εάν και τις μη γεωργικές ενδείξεις αν θα τις καλύψουμε με την ίδια διάταξη. Ε, φυσικά δεν είναι δυνατόν η σαμπάνια ε, να πούμε ότι δεν μπορεί να βγει πέραν της ε, καμπανίας διότι είναι αλλιώς το κλίμα και το έδαφος. Ξέρει τις θέσεις μας πάντως η συγκίτρια και ξέρει ότι αυτή την τροπολογία δεν θα την ψηφίσουμε. Άρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου συνολικά. Θεωρώ ότι πετύχαμε αξιόλογη συμφωνία και θα δώσουμε πράσινο φως στο κείμενο. Ευχαριστούμε κύριε Ντάλτον, λέει ο Πρόεδρος, για την άλλη τώρα. Ο κύριος Γκουόγκα. Σας ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την ε, επικοδομητική δουλειά, γιατί συνολικά θεωρούμε ότι η γνωμοδότηση είναι καλή και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εισηγητρία και τα πολλά άλλα μέλη που υποστηρίξαν τη διαδικασία. Ωστόσο, έχουμε σημαντικά θέματα με τον 9, 15, 19, 21 και 22. Ιδιαίτερα με αυτούς τους συμβιβασμούς λοιπόν. Και νομίζω ότι με το ΕΣΙΑ και το ΕΛΚ είμαστε ιδιαίτερα σε Συμφωνούμε. Και οι 23 και οι 19, 21, 22 μας προβληματίζουν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξουν. Σε ό,τι αφορά τον γεωποκλεισμό, ο συμβιβασμό ε, είναι πολύ αδύναμο. Θεωρούμε ότι πρέπει να καταθέσουμε μια πιο φιλόδεξη ε, πρόταση. Επίση, ε, η άλλη δεν μπορεί να υποστηρίξει αρνητική διατύπωση για την συνεργατική οικονομία σε τομεί όπω είναι η φορολογία, σε ό,τι αφορά την συνεργατική οικονομία. Θα την υποστηρίξουμε τη συνεργατική οικονομία. Ούτε το ΜΕΙΔΙΝ μπορούμε να υποστηρίξουμε και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεωρήσει όλε τι προδιαγραφέ για την επισήμανση και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τα πλέον ουσιώδη στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατανάλωση των προϊόντων. Η Άλτα επίση θεωρεί ότι θα πρέπει να δίδεται ε, πληροφόρηση μέσω ψηφιακών μέσων και όχι πάνω στο προϊόν. Και επίσης πιστεύω ότι η 22 λοιπόν, η συμβαστική 22 δεν είναι επαρκώς φιλόδοξη πολύ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο και τώρα δεν έχουμε κανέναν από την ΚΟΕ. Από τους πράσινους είναι η Τζούλια Ρέντα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ο κύριος Ρέντα μάλλον. Ευχαριστώ πολύ θα μιλήσω εκ μέρους της Τζούλια Ρέντα, που είναι σκιώδης για την ομάδα μας. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Έλαβε υπόψη τις απόψεις μας για τη χρηματοδότηση, τη συνεργατική οικονομία, τις προδιαγραφές που μπορούν να εφαρμόζονται εύκολα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ανοιχτά μοντέλα διοδότησης. Είμαστε πολύ θετικοί. Υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες όμως από πλευρά ομάδα μα για τον ε, γεωγραφικό αποκλεισμό, geo-blocking. Ε, πετύχαμε κάποιου συμβιβασμού όσον αφορά τι διαπραγματεύσει στην ψηφιακή αγορά και θα έπρεπε να ληφθούν καλύτερα υπόψη. Δεχόμαστε την ανάγκη για φιλόδοξο στόχο για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, geo-blocking, αναγνωρίζοντα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα υποχρεώνονται να ε, παραδίδουν τι υπηρεσίε του παντού. Πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα δικαιώματα των καταναλωτών για πρόσβαση στι πληροφορίε στα αγαθά, που δεν το ίδιο σαν να υποχρεώνει τι εταιρείε να παραδίδουν παντού τα προϊόντα. Όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, γεωγραφικέ ενδείξει, δεν συμφωνούμε με αυτή την τοποθέτηση. Και όσον αφορά τις εξαιρέσεις και λοιπά και προτιμησιακά καθεστώτα, θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για την ομάδα μας για να τονωθεί η παραγωγή γενοσύμων ε, και παρομοίων φαρμάκων. Έχουμε συγκλίνουσες τροπολογίες ομάδων. Ελπίζουμε ότι θετικό αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι εφικτό. Επ' αυτόν. Η τροπολογία μας 219 ε, ε, και 220 συγκλίνουν αλλά έχουμε προβλήματα με την τροπολογία 220 εκεί που λέει χωρίς να υπονομεύουμε την αγορά που ε, ε, χορηγείται αποκλειστικά μέσω ε, των προτιμησιακών καθεστώτων σε αποκλειστικές αγορές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Άλμπρεχτ. Πάμε στο FTD. Ο Μάρκο Τζούλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια τον, ε, για τη δουλειά που έγινε. Το ξεκινήσαμε από θετικά στοιχεία, το βελτιώσαμε το κείμενο και συμπεριλάβαμε διάφορα στοιχεία. Είναι σημαντικό και το εξή. Στο κείμενο διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα του πολίτη είτε είναι εργαζόμενος είτε καταναλωτής τονίζουμε τη σημασία να έχουμε θετικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε σαφούς, σαφή συγγνώμη και απλούς κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, μας ικανοποιεί η προσέγγιση στην οποία καταλήξαμε για αυτή την οικονομία στη συνεργατική οικονομία θα πρέπει να ζητήσουν τον νομοθέτη να καταβάλει προσπάθειες για να εφαρμοστούν προδιαγραφές που θα λαμβάνουν υπόψη την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το τομέας και κατά κάποιο τρόπο να προβλέψουμε μέσω ευέλικτης νομοθεσίας τη δυνατότητα να καλύψουμε νέες ανάγκες απασχόλησης και θέσεις εργασίας που ακόμα δεν έχουμε υπόψη μας ποιες μπορεί να είναι. Μας πει το αίτημα για νομοθετική παρέμβαση υπέρ των γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που δεν είναι αγροτροφημικά. Αυτό δεν αντιβαίνει την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων, αντιθέτως επιτρέπει την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στην Ήπειρό μας. Εξίσου υποστηρίζουμε την τι πληροφορίε που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι πληροφορίε που θα δίδονται για την προέλευση των προϊόντων, τι θα αναφέρει η ετικέτα. Αυτό είναι άλλο ένα σύστημα που δίνει περισσότερε πληροφορίε στον καταναλωτή. Έτσι ο καταναλωτή μπορεί να κάνει επιλογέ καλύτερα ενημερωμένο. Άρα αυτό δίνει προστιθέμενη αξία. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τη δυνατότητα παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη ε, πριν να λήξει άδεια Εκεί δεν έχουν πετύχει καλό συμβιβασμό. Εγώ και άλλοι συνάδελφοι υποβάλαμε σχετικές τροπολογίες και ελπίζουμε αυτές να υπερψηφιστούν διότι διαφυλάσσεται το δικαίωμα των κατόχων Αδίες και αυτό επιτρέπει στην Ήπειρο να έχουμε κύκλο παραγωγής ε, να υπάρχουν κύκλοι παραγωγής που τώρα βρίσκονται σε τρίτες χώρες και ελπίζουμε τελικά να υπάρξει θετική προσέγγιση όσον αφορά τις τοπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Τζούλου. Δεν βλέπω άλλους να θέλουν πάρει το λόγο. Από πλευρά ομάδων θα δώσω το λόγο στους άλλους βουλευτές. Συνάδελφε ΣΒΑΜ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Ιταλίδα συνάδελφο, για την εξαιρετική πραγματικά δουλειά που έκανε, γιατί πιστεύω ότι το κεντρικό μήνυμα το οποίο απορρέει από την έκθεση αυτή πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εστιαστεί στο ότι ω Κοινοβούλιο ε, για την εφαρμογή και την καλύτερη ε, εφαρμογή των ε, προδιαγραφών της ε, οδηγίας για την ιστορική αγορά υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι υπάρχει αυτή η βασική γραμμή για όλους τους πολίτες από όπου και αν προέρχονται και ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ε, θα πρέπει να υποστηρίξει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Το, η έκθεση αυτή νομίζω θα πρέπει να καλύπτει και πολλούς πολιτικούς τομείς. Υπάρχουν και συμβιβασμοί οι οποίοι έχουν επιτευχθεί. Ε, ο συνάδελφος από τους πράσινους επεσήμανε τι γίνεται με τον τομέα των γενοσύμων, ότι είναι σημαντικό ο τομέα αυτό για αυτού ε, και φυσικά τίθεται και το θέμα του περιβαλλοντικού κλάδου, είναι θέμα αρμοδιότητα και του και τη ε, Επιτροπή Περιβάλλοντο. Οπότε ενδεχομένω τα πράγματα να μην είναι ακριβώ όπω τα έχει εφάσιστεί. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο συναδελφό Γκουόγκα μίλησε για το τομέα τη ε, χώρα προέλευση, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται, πρέπει να σας πω ότι και στο σκόλπους του ΕΛΚ τα συζητάμε με επικριτική διάθεση και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Επίτροπο με την υποστήριξη και τη εισηγήτρια και των υπόλοιπων συναδέλφων και ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σφάπ και τώρα η κυρία Γκράφη έχει το λόγο. Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να α, ευχαριστήσω την κυρία Κόμη, την εισηγήτρια και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Μαρλέν γιατί αποδέχτηκαν την ε, πρόσκληση της ε, ομάδας για το PMO και πολλοί που συμμετείχαν ε, στην ομάδα ανέφεραν ποια ήταν η θέση τους για την έκθεση και εκτιμήσαμε λοιπόν την ανταλλαγή αυτή απόψεων με τους ε, συμμετέχοντες, τους πορείς της αγοράς. Θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι γιατί 20 από τις τροπολογίες μου ε, συμπεριλήφθησαν στους συμβιβασμούς. Ωστόσο, 8 δεν συμπεριλήφθησαν, αλλά όλες αυτές οι τροπολογίες ε, ως σκοπό έχουν να ε, συνδράμουν και να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα θέλαμε να δώσουμε μία πνοή στην αγορά με την έκθεση αυτή, να υπάρχουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να καλέσω καλέσετε τον κύριο Ντάλτον για ένα καφέ για να του εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο η σαμπάνια που προστατεύεται από τη γεωγραφική ένδειξη, αλλά υπάρχουν και άλλα προϊόντα, όπως τα κεραμικά, για παράδειγμα, τα οποία επίσης ε, προστατεύονται γιατί για παράδειγμα τα κλαμβάνουν άργυλα όπως συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε βασικά, να συνδράμουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των ε, μικρομεσαίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχουν ζητήσει άλλη το λόγο και άρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Όσον αφορά κυρία Μίτση, εισηγείται τη ομάδα, νομίζω ότι είναι ισορροπημένο το κείμενο, κυρίω όσον αφορά του συμβιβασμού. Ελπίζω να τύχει υποστηρίξεω μεγάλη, διότι η ισορροπία βρίσκεται με κοινή προσπάθεια. Όλοι να προσπαθούμε να περάσουμε κάποια στοιχεία και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Θεωρώ ότι κινούμε θα σωστή κατεύθυνση σαν Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή. Όσον αφορά το made in, ε, τις γεωγραφικές ενδείξεις και ε, την αναφορά κατασκευής του προϊόντος, παραγωγής του προϊόντος. Υπήρξε ευρία υποστήριξη. Αύριο θα ψηφίσουμε. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα θα ψηφίσουμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κόμη να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο διευκρινήσεις να κάνω. Λοιπόν, η πρώτη όσον αφορά το σύστημα των φαρμάκων, όπως είπαμε, σε διάφορες συναντήσεις. Δεν θέλησα να εμβαθύνω στο θέμα, διότι θα καταφτάσει μελέτη συνεπιών αντικτύπου για αυτό το θέμα και για τα γενώσιμα και για τα λοιπά πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν θα έχουμε το κείμενο αυτό, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ζητούν οι πολίτες, τι ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτές που παράγουν τα γενώσιμα και αυτές που παράγουν τα άλλα φάρμακα. Εν αναμονή του εγγράφου ενισχύσαμε έτσι περαιτέρω το σύστημα των ευρεσιτεχνιών, των αδειών, διότι λειτουργεί άριστα σε όλα τα κράτη-μέλη. Κυρίως η χρόνη προστασία, το χρονικό διάστημα προστασίας. Τώρα, τις ενδείξει προελεύσεως και που έχουν παρασκευαστεί τα προϊόντα, αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, το έχω συνηθίσει στη συζήτηση σε σχέση με τις προηγούμενες, φορά, προηγούμενες φορές έχουμε μελέτη συνεπειών που καθόρισε τη σημασία των ενδείξεων προελεύσεως για τους καταναλωτές. Λοιπόν, αναλύσαμε ε, τα πράγματα διαφορετική σκοπιά. Τα προηγούμενα χρόνια πάντα θεωρούσαμε ότι η ένδειξη αυτή προελεύσεως ήταν υπέρ της επιχείρησης ή της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αντίθετα, από τη μελέτη συνεπιών που ρωτήσαμε την άποψη των καταναλωτών, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να κατακαιρματίσουμε και να διαιρέσουμε έτσι περαιτέρω την αγορά. Αντιθέτως θέλουμε αυτό που είναι και ο τίτλος της επιτροπής μας. Θέλουμε να πετύχουμε την προστασία των καταναλωτών εντός της αγοράς. Δεν ξέρω τι κακό έχει να λέμε ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε σε μια χώρα και όχι σε άλλη. Δίνει κάποια αξία στο ίδιο το προϊόν. Και μπορεί ελεύθερα ο καταναλωτής μετά τι θα αγοράσει, πώς θα ξοδέψει τα χρήματά του. Ευχαριστώ πολύ όλους. Θα ψηφίσουμε αύριο. Ελπίζω όλοι μαζί να πετύχουμε την καλύτερη συνένεση, διότι είναι ε, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει γρήγορα στην Επιτροπή για να δοθούν κατάλληλες απαντήσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο. υπηρεσίες. Η Λούση Άντερσον είναι η συγκίτρια αυτής της έκθεσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά μου και ευχαριστώ και όλους τους ε, σκιώδες εισηγητές. Και είχαμε και χθες πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην ε, αρμόδια ομάδα και επίσης ευχαριστώ και όλους όσους υπέβαλαν κάποιες τροπολογίες. Συνολικά έχουμε 53 από όλες τις πολιτικές ομάδες. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης είχαμε μια σειρά ζητημάτων σημαντικών τα οποία ανεδίθησαν από αυτές τις τροπολογίες και έτσι τώρα έχουμε μια πληρέστερη έκθεση και θα πρέπει να ε, αγκαλιάσουμε όσο γίνεται περισσότερες και όσο γίνεται περισσότερα θέματα και όλα αυτά κατά τρόπο έφτακτο. Τώρα κάτι άλλο. Ε, θέλουμε τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την, την οδηγία ε, και ευέλικτα, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν ορθά. Και αυτό προκύπτει από πολλές τροπολογίες. Τώρα, αυτού τις καθολικές υπηρεσίες, το αν είναι βιώσιμες, θα εξαρτηθεί από τα κράτη-μέλη. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφορές αν θα πρέπει κανείς να χτενίσει την νομοθεσία. Πάντως ε, όλοι υπέβαλαν στις τροπολογίες και επίσης έχουμε ε, μνήα στο θέμα της παράδοσης δεμάτων της σχετικής υπηρεσίας λοιπόν και επίσης υπάρχει ευρεία συνέντευξη ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να κάνει όσον αφορά, νουλάνε και η αυξανόμενη παράδοση δεμάτων διασυνοριακά θα πρέπει να έχει καλές τιμές, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυτό να εξυπηρετεί επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Επίσης είπαμε τα της ε, αποζημίωσης των ε, καταναλωτών ε, για κάποιες μικροαξιώσεις, επίσης ότι θα πρέπει κάποια μέλη, κράτη-μέλη να μεταφέρουν πλήρως και σωστά την οδηγία ADR για την αποζημίωση των καταναλωτών και επίσης αναφέρθηκαν και οι εργαζόμενοι και είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει βιωσιμότητα γενικά σε αυτόν τον ε, τομέα ε, για παιδεία, κατάρτιση και γενικότερα ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Επίσης είπαμε τι θα γίνει ε, με τους φραγμούς στην προσβασιμότητα νέων παικτών ή νέων παρόχων και είπαμε ότι Έχουμε ένα αρχικό κείμενο αυτών των συμβαστικών. Ε, διανεμηθεί χθε. Έγινε μια πολύ καλή συνεδρίαση των σκιωδών ή εισηγητών και θα το επεξεργαστούμε κι άλλο τα θέματα γιατί μπορεί να προκύψουν κι άλλε συμβαστικέ πρωτοβουλίε. Για άλλη μια φορά να σα ευχαριστήσω. Είναι πολύ σημαντικός ο κλάδο αυτός και νομίζω ότι βόηθησε και η Επιτροπή. Ευχαριστούμε η Ευχαριστούμε την κυρία Άντερσον και τώρα σκιώδες εισηγητές. Η Ρόζα για το ΕΛΚ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πολύ τη Λούση για τη δουλειά που έκανε. Το θέμα είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό και αυτό γιατί οι ταχυδραμικές αυτές οι υπηρεσίες όπως ξέρουμε επηρεάζουν πάρα πολύ την ιστορική αγορά και φυσικά την ψηφιακή διάσταση. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουμε και να φροντίσουμε να λειτουργεί σωστά. Διάβασα λοιπόν το σχέδιο της έκθεσης της Λούση. Ε, είναι πάρα πολύ καλό. Αποτελεί μια πολύ καλή, καλό σημείο κίνησης για την, ε, τη συζήτηση. Καταρχά, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, οι στόχοι της οδηγίας, όπως είναι για παράδειγμα να επιτευχθεί μια ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά ε, τις υπηρεσίε υπηρεσίες έχουν επιτευχθεί. Δεν το πιστεύω. Έχουμε 28 διαφορετικές αγορές από ό,τι ξέρετε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα Κατακαιρματισμό. Και το έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθολική υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ε, εφαρμόζεται με πολύ ξεχωριστό τρόπο σε κάθε κράτος μέρο και δεν ε, εγγυάται σαφήνεια. Αλλά αυτέ οι 28 αγορές έχουν ένα πράγμα κοινό. Όλοι πιστεύουν, όλοι οι παροχοί σκέφτονται εντό του πλαισίου της χώρας τους και πιστεύω ότι δεν μπορούν τα σύνορα να αποτελούν φραγμό και όριο θα πρέπει να σημαίνουν τα σύνορα επιπλέον κόστος. Δεύτερο ζήτημα είναι φυσικά το θέμα της εφαρμογής. Η Κομισιόν έδωσε πάρα πολύ χρόνο στα κρατημέλη να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία. Δύο χρόνια σχεδόν περίμενε. μετά την προθεσμία που οριζόταν στην οδηγία για την, εφαρμογή, τη δημοσίευση της έκθεσης. Δυστυχώ αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα εφαρμογή. Έχουμε δύο διαδικασίε παραβάση που έχουν ξεκινήσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τότε το αντικείμενο τη ε, εφαρμογή στα κράτη-μέλη είναι σαφέ ότι συχνά δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή. Υπάρχουν θέματα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό των δομών, σε ό,τι αφορά τι ρυθμιστικές ε, υποδομές, θέματα κατοχής, έλεγχου, αλλά πάνω από όλα υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια για τους ε, παρόχους σε ό,τι αφορά την πρόσβασή στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν από όλων αυτών να εξκύψουμε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις υποδομές, αλλά μέχρι και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ως σκοπό έχουν να προστατεύσουν τους εσωτερικούς ε, παρόχους. Άρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι 11 κράτη-μέλη φαίνεται ότι έχουν όρους ε, αδειοδότησης που ουσιαστικά επαναλαμβάνουν διατάξεις άλλων νομοθετημάτων. Δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ υπερβολικά σε θέματα εφαρμογής, αλλά θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Τρίτο σημείο τώρα. Εμεί είμαστε, θεωρώ, η Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για θέματα ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, να δώσουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική σε ό,τι αφορά την παράδοση πακέτων. Να δούμε ότι η αναποτελεσματικότητα της αγοράς αυτής τελικά ε, θα κάνει τις ε, επιχειρήσεις ε, online να γίνουν και αυτή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών για παράδοση πακέτων. Ε, η Amazon, για παράδειγμα, πριν από κάποιε εβδομάδε, μάθαμε ότι θα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα έχει κάποιε δυνατότητε για παράδοση πακέτων. Δεν είναι απειλή αυτό, βέβαια, αλλά θα προτιμούσα να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο την αγορά αυτή. Θα ήθελα να συζητήσουμε διάφορα καθεστώτα ε, σε ό,τι αφορά το οργανωτικό σκέλος που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Θα ήθελα επίσης ε, να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα ταχυδρομικά πακέτα, τι γίνεται με τα πακέτα που παραδίδονται Και Λούση, λοιπόν, με χαρά θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σου, να θέτω τα ρήματα αυτά, ε, να ψάχνουμε απαντήσεις και ίσως να αναζητούμε και εντελώ νέες λύσεις. σε ό,τι αφορά και την ομάδα εργασία, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβασης. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε καινούριε ιδέε. και πραγματικά έχει έρθει η ώρα να βελτιώσουμε την κατάσταση. για την αγορά αυτή η οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά παροχημένη. Σε ευχαριστώ κύρια Τούν. Τσέζακ για το ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τη Λούση Άντερσον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Κιώδης, οι οποίοι επεξεργάστηκαν το θέμα μαζί της. Εξέτασα τις συμβαστικές λύσεις που ετοιμάστηκαν και θα ήθελα να εκφράσω τι ευχαριστίε μου που συμπεριελήφθησαν οι δικές μου τροπολογίες στις συμβαστικές που προτείνονται. Κυρίως εκείνες οι οποίες, οι οποίες λέγω αφορούσαν την ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις νοριακές υπηρεσίες. Δεν έχω άλλα συγκεκριμένα σχόλια. Όμως θα ήθελα να πω και το εξής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγγυηθεί τις καλές συνθήκες εργασίας, μάλλον ζητά να επικρατούν καλές συνθήκες εργασίας για εκείνους που εργάζονται στα ταχυδρομεία. Πολύ το προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπαίνει στα χωράφια ε, των κρατών μελών. Πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτά πρέπει να είναι υπεύθυνα για αυτό το ζήτημα και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζω ότι θα γίνει κι άλλη δουλειά όσον αφορά τη γνωμοδότηση και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιους συμβιβασμός και στο θέμα που μόλις σας επισήμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσέζακ. Γκάρντ για την Άλντε. Συνάδελφοι έχετε το λόγο. Ο κύριος Γκάρντ, ευχαριστώ. Και από πλευράς φιλελευθέρων θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εμείς την εισηγήτρια. Πολύ καλή δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Ήδη στις δύο συναντήσεις που συμμετείχα διαπίστωσα ότι υπήρχε καλή θέληση και συνεργατικό πνεύμα επικράτησε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον η ομάδα των φιλελευθέρων ακολουθεί την ίδια προσέγγιση όπως το ΕΛΚ. Νομίζω ότι η κυρία Τούν ήδη είπε σωστά πράγματα, πολύ συνετά, πρέπει να εστιαστούμε επί της αγοράς, πώς λειτουργεί αυτή, που έχει προβλήματα στον αφορά τη λειτουργία της σε πολλά κράτη-μέλη. Με την έκθεση πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους άλλους και στα κράτη-μέλη ότι θέλουμε να λειτουργεί καλύτερα η αγορά. Άλλο θετικό σημείο από αυτά που έθεσε η κυρία Τούν είναι και το εξή. Ίσως θα έπρεπε να υποβάλουμε μία-δύο τροπολογίες σχετικά με το μέλλον. Το μέλλον του τομέα πήγα στις ΗΠΑ. Με την Επιτροπή Απασχόλησης θέλαμε να δούμε την Amazon και τις άλλες εταιρείες πώς λειτουργούν μπορείτε να έχετε πολλές απόψεις για τις εταιρείες αυτές και πώς λειτουργούν. Αν τις δεις από την πλευρά των εργαζομένων, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το μέλλον. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν συζητούμε τις δικές μας αγορές και τις δικές μας ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ίσως το μέλλον θα πρέπει κάπως να αντικατοπτρίζεται. Δεν το συζητήσαμε στην πρώτερη συζήτησή μας, αλλά μου έρχεται στο μυαλό ότι ίσως αυτή είναι καλή ιδέα να σκεφτούμε και ποιο θα είναι το μέλλον της αγοράς αυτής και κάτι να αναφέρουμε στις τροπολογίες. Δεν θα χρονοτριβήσω, θα ήθελα να πω ότι παρακολουθούμε την κατεύθυνση που ακολουθεί και το ΕΛΚ, συμφωνούμε με την προσέγγιση του ΕΛΚ. Και η συγγήτρια έδειξε πολύ καλή θέληση και νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια αξιοπρεπή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ευχαριστώ κύριε Λόκεργαρτ. Δεν έχουμε άλλους σκιώδεις εισηγητές, δεν έχουμε εκπροσώπους των άλλων ομάδων παρόντες, λοιπόν. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Λούση αν θέλει να απαντήσει. Ορίστε Λούση. Ευχαριστώ για τις χρήσιμες παρατηρήσεις που προσθέτουν στα όσα ήδη συζητήσαμε. Ρόζα έχει 100% δίκιο όσον φορά την ψηφιακή πτυχή. Εν μέρει τα συζητήσαμε και νομίζω θα το πετύχουμε. Επίσης όσον αφορά την ε, μεταφορά του κειμένου, όσον αφορά του στόχους μας, θα πρέπει να δούμε πώς θα τους τακτοποιήσουμε αυτούς τους συμβασμούς, τόσο ώστε να πιάσουν τόπο περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι κανεί ρίχνει το βάρο στο τι γίνεται στο ιστορικό κάθε κράτο μέλο και όχι διασυνοριακά. Αλλά εμεί δεν το ρίχνουμε αυτό. Κανεί άλλο δεν το κάνει πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Αλλά και για το στοιχείο του μακροπρόθεσμου και για την υποχρέωση ε, δυνατότητας πρόσβασης. Το θέμα των εργαζομένων είναι σημαντικό, αλλά θα βρεθεί κάποια λύση και έτσι θα ρυθμιστεί το θέμα του ποιος φέρει την ευθύνη. Ε, να δούμε και αυτό το οποίο είπαν οι φιλελεύθεροι για την αγορά και εμείς όπως και άλλες πολιτικές ομάδες. Θεωρούμε ότι έτσι πιθανώς θα λειτουργεί καλύτερα η ενιαία αγορά. Τώρα όσον αφορά την Amazon και της είπα, με τίποτα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις εξελίξεις. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ε, με κάποιο συντεταγμένο και αξιοπρεπή τρόπο γιατί αυτό θα είναι προς το όφελος όλων. Βεβαίως και πρέπει να γνωρίσουμε τις ε, εξελίξεις αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να κάνουμε το σωστό. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Άντερσον. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα. Thank you, Mr. Uh, all. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που συμμετείχαμε σε αυτή τη συζήτηση και χαιρόμαστε που το θέμα αυτό προσελκύει πολύ μεγάλη προσοχή από πλευρά τη ε, Επιτροπή σα, γιατί απασχολεί και του πολίτε. Ε, δύο-τρία θέματα τώρα σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή που είπε και η Λούση. Συμφωνώ με αυτά που είπε για τη σωστή εφαρμογή σε ό,τι αφορά τη σημασία, για παράδειγμα, ε, των ταχυδρομικών πακέτων. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά θέματα. Η κυρία Τούν έφτασε το θέμα του κατά πόσον ο στόχο της οδηγία έχει επιτευχθεί. Και είπατε ότι ο βασικός σκοπός ήταν η ενιαία αγορά. Σε κάποιο βαθμό συμφωνώ. Θα ήθελα να σας πω ότι τότε είχαμε πει ότι δύο είναι οι βασικοί σκοποί. Καταρχά, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματο, η ποιότητα του συστήματο, η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και εκ παραλλήλου η αποδοτικότητα προ το κέρδος γιατί όταν ξεκινήσαμε ήταν δύο μόνο υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ήταν ε, κερδοφόροι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει Άρα, σκοπό είχαμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και το κερδοφορία, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος των κοινοφελών υπηρεσιών. Το πετύχαμε λοιπόν και αυτό τον δεύτερο στόχο. Παρέχονται οι καθολικές ε, κοινοφελείς υπηρεσίες και, και στο θέμα της ανταγωνιστικότητα ενδεχομένως να μην πετύχαμε τόσο καλά και αυτό γιατί όπως και εσείς είπατε η μεταφορά, η εφαρμογή δεν ήταν τόσο φιλόδοξη όσο θα θέλαμε. Ήταν λοιπόν πάντα εύκολη η εισαγωγή στην αγορά και όταν έτυχε διαπραγματεύσει η τρίτη οδηγία ήταν σε αυξητική τάση η αγορά, ενώ τώρα είναι σε πτωτική τάση. Ο τρίτο σκοπό ήταν η ανιαία αγορά. Αλλά αυτό ήταν λιγότερο μεγάλο ζήτημα για σήμερα όμως και τώρα στι σημερινές ανάγκες. Βλέπουμε το τι θέλουν και τι χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Κυρίω πακέτα και λιγότερο γράμματα. Και τα πακέτα γίνονται όλο και πιο πολύ μεγάλο θέμα γιατί με τη συνδυασμό των θεμάτων όπως ο γεωποκλεισμός, αν θέλει κανείς να μεγαλώσει η επιχείρησή του και να ε, επεκταθεί και διασυνοριακά χωρίς μια σωστή παροχή ε, και παράδοση πακέτων δεν μπορεί να το πράξει. Αυτός ε, λοιπόν είναι, την νέα κατάσταση και πρέπει να πούμε ότι έχουν αλλάξει και κάπως οι στόχοι μας επειδή έχει αλλάξει και η αγορά σε ό,τι αφορά θέματα εφαρμογή τώρα καθε αυτής. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε την αίσθηση ότι κάποια κράτη-μέλη ενδεχομένω να μην έχουν επιδείξει τον ε, ενθουσιασμό που θα θέλαμε να δούμε σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της αγοράς και εκ παραλλήλου η εφαρμογή πάντα είναι θέμα δύσκολο γιατί η οδηγία αποτελεί μια οδηγία πλαίσιο γενικών γραμμών που αφήνει μεγάλο περιθώριο λιγμού για τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε λοιπόν να δουλέψει αυτό, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν μαζί μας και για τους στόχους. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να διακόσουμε να αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να προβαίνουν σε ενέργειες που δεν επιθυμούν. Η ενιαία αγορά λοιπόν δεν είναι έτσι, οι θα πρέπει να είναι παντού. Κύριε Τσεσάκα και συγγνώμη γιατί δεν προφέρω στο όνομά σα λέει ο μιλητή. είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγυάται καλέ ε, εργασιακέ συνθήκε και ότι το παρακάναμε και θα πρέπει να αυτό να μείνει ω αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αν δεν παρανόησα αυτά που υπόθηκαν, δεν το κάναμε αυτό. Αποτελεί αυτό αρμοδιότητα των κρατών μελών και το αναγνωρίζουμε σε όλη την οδηγία. Οι κοινωνικέ συνθήκε, οι εργασιακέ συνθήκε, σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, όλα αυτά γίνονται βάσει εθνική νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθήσαμε, δεν επιχειρήσαμε να μπούμε στα χωράφια των εργασιακών συνθήκων. Ο κ. Λόκγκαρτ αναφέρθηκε στην ανάγκη να λειτουργούν καλύτερα οι αγορέ. Είδα και τι τροπολογίε σα, τι αναφορέ που κάνατε στα ποσοστά των εργαζομένων και ούτω καθεξή. Κοιτώντα τι γίνεται στη Δανία, στην αγορά εργασία, είναι η πιο ακραία περίπτωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο λόγω των πολιτών που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μίδια και στέλνουν ε, mail, οι επιχειρήσεις στέλνουν ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πιο πολύ ε, ηλεκτρονικά μέσα. Και έτσι λοιπόν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ταχυδρομείο μάλλον στην Δανία, είναι στο 40% των ε, τον που είχε πριν από κάποια χρόνια. Και εξακολουθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα νομικό περιβάλλον το οποίο ορίστηκε σε άλλες εποχές. Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο θα πρέπει από κοινού να κάτσουν να σκεφτούν το τι θα συμβεί σε 5-10 χρόνια, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μεγιστοποιήσει τα ωφέλη για τους πολίτες, τους φορολογούμενους και καθεξής. Κάναμε και μία τέτοια σχετική συζήτηση πριν από κάποιες εβδομάδες και η Ελλαδική Προεδρία ρώτησε τα κράτη-μέλη κατά πόσον βάσει της έκθεσης αυτέ πιστεύουν ότι το τρέχον πλαίσιο να εξακολουθεί να εξυπηρετεί το σκοπό τους και ότι είναι αρκετά ευέλικτο και κατά πόσο αυτό θα ισχύει σε 5-10 χρόνια. Σήμερα λοιπόν τα πιο πολλά κράτη-μέλη δηλώνουν ότι ε, τα βγάζουμε πέρα. Κακήν κακό, λίγο πολύ με κάποιε λύσει. αλλά σχεδόν όλα τα κρατημέλη στην αίθουσα συμφώνησαν ότι σε 5-10 χρόνια ενδεχομένως να χρειαζόμαστε κάτι καινούριο. Άρα αυτό μα απασχολεί όλου. Θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι θα χρειαζόμαστε, τι θα χρειαζόμαστε και τι θα χρειάζονται και οι πολίτε μα σε 5-10 χρόνια και αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. So I believe we can now move on to the next item. Πάμε παρακάτω, λέει η κυρία Βίκη Φόρτ που ανέλαβε την Προεδρία. Which is the... Και είναι το θέμα υπαριθμών 9 που είναι ανταλλαγή ε, απόψεων όσον αφορά την οδηγία για το νημερωτικό δελτίο. Well, I'm the rapporteur, but if it's okay, I'll just stay in the chair because we're Λίγα λεπτά και μόνο θα σας απασχολήσω, οπότε κρατάω την Προεδρία. Πρόκειται για αυτή την νομοδότηση που θα πρέπει να μας απασχολήσει ως συναρμόδια μαζί με την ΕΚΟΝ όταν αφορά αυτή την, αυτό το, την υποχρέωση του ημερωτικού δελτίου. Στην προηγούμενη εντολή επίσης είχαμε ασχοληθεί, ήμουν ασκιώδης για την ΕΚΟΝ και ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι συγκεκριμένα να σας πω πώς ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται και θα πρέπει επίσης να ε, ε, ε οι ίδιοι καταναλωτέ την πρόσθεση τους. Και τα είπαμε αυτά και με τον κύριο Ντεμπάκερ στην Οικονομική Επιτροπή. Και ό,τι όμως έχει επιπτώσεις για τους καταναλωτές θα έπρεπε να έρχεται σε εμά. Έχουμε υποβάλει 21 τροπολογίες. Πρώτα πρώτα για την περίληψη του δελτίου να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες και είπαμε ότι ε, μόνο σε επενδυτές λιανικής ισχύει αυτό το δελτίο τότε είναι υποχρεωτικό η περίληψη συγγνώμη είναι υποχρεωτική Αλλιώ αν δεν πρόκειται περί ηλιανική τραπεζικής συναλλαγή δεν επιβάλλεται. Ε, είναι και κάτι δαπανηρό. Είπαμε, είπαμε να, δούμε, να ορίσουμε πόσε σελίδε θα είναι, πόσο ε, θα το, μεγάλο το κείμενο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι σωστό πάντων να έχουμε μία λύση για κάθε περίπτωση, οπότε προσπάθησα να, να βάλω πινελιές ευελιξίες και επίση το είπαμε η εισαγωγική σύνοψη ή περίληψη. Αυτό το προσπέκτος τέλο πάντων. Και υπάρχει μια άλλη τροπολογία η οποία μιλά περί μεταφράσεως. Άρα να έχουμε κείμενο σε μια επίσημη χώρα ε, του κράτους μέλους αλλά και να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της οδηγίας PRIPS. Οπότε έτσι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, επενδυτές λιανικών συναλλαγών σε σχέση με ομόλογα χρέους τα οποία εκδίδονται γιατί θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα σε διαφορετικές πηγές πόρων ή κεφαλαίου έχουμε βάλει όριο για αυτά τα ομόλογα τα 100.000 ευρώ και επομένω κάτω από τα 100.000 ευρώ που είναι οι συναλλαγές λιανικής retail banking εκεί θα έχουμε αυτό το φιλικό στον επενδυτή μέτρο της ε, σύνοψης επίσης προτάθηκε να έχουμε πιο επίκη κατόφλια και οροφές για τις ε, μέσου μεγέθους εταιρείε να έχουν πρόσβαση στην κεφαλή αγορά και εγώ θεωρώ προσωπικά ότι τούτο είναι πολύ θετικό και βοηθά τις μικρότερες εταιρείε ούτω ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγορές οπότε και προσωπικά πρεσβεύω ότι θα πρέπει αυτές τις τροπολογίες της ΕΚΟΝ να τις εγκρίνουμε. Αλλά βέβαια θέλω ε, και αυτό να το παληθεύσω σε συζήτηση μαζί σας για τον καταναλωτή. Αυτά από τον κύριο Ντεμπάκερ. Πάντως έχουμε για τα θέματα της δευτερογενούς εκδόσεως ομολόγων. Έχει βάλει εδώ κάποια μήνυμα η Επιτροπή για ε, κάλυψη 70% της έκδοσης ομολόγων και ε, εδώ είναι θέμα το πώς θα εξοικονομηθούν κάποιες δαπάνες και αντιστοίχω και εδώ σε κάποιες ορισμένες μόνο περιπτώσεις επιβάλλεται να υπάρχει αυτή η, η, ε, η, περίληψη. Οπότε έχουμε και εδώ τον, τον ε, του, του, του διαδικτυα, του έρανου αυτού, τη, της συμμετοχής χρηματοδότησης, το crowdfunding. Όμως, έχουμε εδώ πέρα πολλές πλατφόρμες ε, που μπορούν να είναι η αφετηρία της παροχής αυτών των πληροφοριών προς τους καταναλωτάς. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι σαφείς οι πληροφορίες εξού και το υποχρεωτικό. Άρα θα πρέπει να το επεξεργαστούμε κι άλλο το ζήτημα αυτό και γι' αυτό και έχω υποβάλει μια τροπολογία ε, σαν ταξιδιωτική οδηγία φανταστείτε υπέρ του καταναλωτή σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες, τις, τις βάσεις αφετηρίας για το crowdfunding, την χρηματοδότηση με έραν. Ευχαριστώ, Βίκη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτάσεις αυτές. Επαναλαμβάνονται κάποιες προτάσεις τις οποίες μπορούμε να παραδεχτούμε ως έλικα και οι οποίες θα πρέπει να ευχαριστούν στην Επιτροπή ΕΜΚΟ. Καταρχάς, τροπολογία 1 για το crowdfunding. πρόταση 2 σε ό,τι αφορά τα ποσά πάνω από 100.000 ευρώ και τροπολογίες 4, 3, 4 και 5 για το πεδίο εφαρμογή τη πρόταση οδηγία. Και η προσθήκη του μικρού επενδυτή ορισμός στη τροπολογία 6 δεν μας προβληματίσει και ο περιορισμό από πλευρά τη Επιτροπή σε έξι σελίδε και ο περιορισμό των ε, παραγόντων κινδύνου. Αυτά τα θεωρώ προβληματικά. Μάλλον είναι προβληματικά. Σε ό,τι αφορά τα 20 δισεκατομμύρια, τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, αυτό το θεωρώ προβληματικό. Δεν έχει νόημα, πιστεύω. Θα ήθελα να αποφύγω οι επένδυτες ε, σε κάθε κράτος μέλος να έχουν διαφορετικό ε, το όριο ανά χώρα. Αυτό θα προωθούσε τον ε, ενιαίο χαρακτήρα. Επίσης, ε, η τροπολογία 8 για την αναφορά στο χειρότερο σενάριο. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί κάθε ε, καθένας θα μπορούσε να πτωχεύσει και έτσι να ακυρωθεί η αξία του αξιογράφου. Αυτό το ξέρει όμω κάθε επενδυτή. Δεν είναι ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό ως ε, εισαγωγική σύνοψη, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τους παραγόντες κινδύνους, η αξιολόγηση του κινδύνου βάσει πιθανότητων. Πιστεύω ότι μάλλον είμαι επικριτικός γιατί έχει μεγάλες συνέπειες και σε ό,τι αφορά την μετάφραση της ε, σύνοψης είναι καλό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αφήνει στην ευχαίρεια των κρατών μελών για την διεξαγωγή μη της μετάφρασης, αλλά αναρωτιέμαι αν χρειάζεται καν μια τέτοια μετάφραση, γιατί πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν εμπειρία στον τομέα αυτό και τα έγγραφα αυτά είναι ήδη γραμμένα στην συνηθισμένη γλώσσα για τα θέματα αυτά. Άρα η μετάφραση ουσιαστικά μου φαίνεται περιττή για άτομα εκείνα τα οποία είναι ειδικοί για τέτοια θέματα, αφήστε που συνδέεται και με μεγάλο κόστος. Αυτές είναι οι πρώτες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες και χαίρομαι ιδιαίτερος που θα κάνουμε και τις συναντήσεις των σκιωδών για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ωραία, Κραπίνη. Κυρία Κραπίνη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως Είμαι πεπισμένη ότι η συνεργασία μας είναι και θα είναι καρποφόρα. Έχουμε ήδη, έχω ήδη 20 τροπολογίες που υπέβαλα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε, βλέπετε, όπως είπατε, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών που θέλουν να αποκτήσουν αυτά τα αξιόγραφα από τις ε, κεφαλαγορές. Είμαι ικανοποιημένη διότι βλέπω ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην ενημέρωση, στις πληροφορίες που θα διατίθενται στους ε, καταναλωτές. Θα πρέπει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαγορές. Χρειάζεται να επικρατούν συνθήκες για δίκαιο ανταγωνισμό, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Γι' αυτό στις ε, τροπολογίες μου ανέφερα κάποιες πτυχές που θεώρησα σημαντικές, πολύ σημαντικές, κάποιες προθεσμίες σχετικά με το έγγραφο, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες που χορηγούνται στον καταναλωτή. Πιστεύω για να πετύχουμε την αναγκαία αμεροληψία στο σημείο 58 του κειμένου που λέει ότι υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που καθορίζονται ούτως ώστε εκείνος που εκδίδει τα αξιόγραφα να μπορεί να δημοσιεύει το περιεχόμενο αυτών Πιστεύω ότι αυτή η περίοδος θα πρέπει να ισούται με το χρόνο που δίνουμε στον επενδυτή για να μπορεί να, αξιοποιήσει, να αξιολογήσει την προσφορά και ενδεχομένως να αποσύρει το ενδιαφέρον του αν το επιθυμεί για τα αξιόγραφα. Θα ήθελα στην ομάδα να το συζητήσουμε το θέμα. Έχω υποβάλει 20 τροπολογίες όπως προανέφερα. Δεν κατάλαβα πολύ καλά γιατί χρειαστήκαμε τόσες μέρες. Γιατί θέλαμε 5 συν 10, δηλαδή 15 μέρο, για να συνταχθεί αυτή η γνωμοδότηση, ή μάλλον και να συνταχθεί αυτό το φυλάδιο, το ενημερωτικό. Όλες οι άλλες τροπολογίες επικεντρώνονται επί των φυσικών προσώπων, που είναι και οι πιο ευάλωτοι. Διότι θα μπορούσαν να είναι και καταναλωτέ. Μεταξύ των καταναλωτών έχουμε και πολίτε, όχι απλώ επιχειρήσει. Έχουμε και απλού πολίτε. Θα σα διαβιβάσω τι τροπολογίε μου και περιμένω ακόμη πλευρά των συναδέλφων και άλλε απόψει που θα εκφραστούν στην ομάδα μα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, εναρμόνιση ε, τη δημοσίευση του ενημερωτικού φυλαδίου. Έτσι δημιουργούμε μια νέα αγορά. Ένα, είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς και να γίνει και πιο αποτελεσματική αγορά και οι αγορές εν γέννη. Η εναρμόνιση των κανόνων για το φυλάδιο είναι πολύ σημαντικό σημείο. Οι επενδυτές αποκτούν σαφείς πληροφορίες για να αποφασίσουν για τις επενδύσεις τους. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για τις μικρομέσες επιχειρήσεις, διότι οι κανόνες για το φυλάδιο έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το διοικητικό άχθος και το κόστος να μειωθεί για το φυλάδιο. Κατά την άποψή μου υπάρχουν ένα-δύο σημαντικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν όσον αφορά τον κανονισμό για τα φυλάδια. Ο, το, το το, έχουμε 400.000 ευρώ σαν όριο και ένα εκατομμύριο ανώτατο. Στο άρθρο 3 βλέπουμε ότι τα κρατη μέλη μπορούν να αποφασίσουν για ένα όριο που υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανονισμό ή που υπόκεινται ε, διαδικασίες στον κανονισμό. Μπορούμε με αυτή την προσέγγιση να κατακαιρματίσουμε την ενιαγορά. Εδώ έχουμε έναν κανονισμό και πρέπει να λειτουργεί ως κανονισμός. Άλλο θέμα, η έννοια της σύνοψης που πρέπει να ταιριάζει με το, γενικά με τις οδηγίες για το έγγραφο, για το φυλάδιο. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η σύνοψη πρέπει να αποτελείται μόνο από συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές για τους επενδυτές, ούτως ώστε να μπορούν να αποφασίσουν. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες της σύνοψης. Πιο σημαντικό είναι να πούμε ποια βασικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στο συνοπτικό κείμενο αντί να έχουμε πολύ, πολλές λεπτομέρειες για τους κανόνες. Για να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες χρειάζεται μια πλατφόρμα online. Το ESMA θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα διαδικτυακή. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ψηφιακές για το φυλάδιο αυτό. Θα υποφεληθούν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερη πρόσβαση, πιο εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και αυτές είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανδρέας. Yeah, so Σε ευχαριστούμε, Βίκη, για την ε, πολύ καλά προετοιμασμένη ε, γνωμοδότηση. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Πασκό. Και θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κρίσιμα σημεία σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, γιατί οι κίνδυνοι που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει και των πιθανότητων και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες δεν μπορούν να καταχθούν σωστά. Γιατί οι οικονομικοί κίνδυνοι πολύ απλά δεν μπορούν να μπουν και να συνοψιστούν σε πέντε κατηγορίες και μετά να θεωρούμε ότι είναι εύκολα κατανοητοί Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην δημιουργούμε λανθασμένε εντυπώσεις κατά δεύτερον, Πρόεδρε. Το είπε και ο συνάδελφος Αριμό. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί θα πρέπει να καταργηθεί η σχετική, ε, οι σχετικές υποχρεώσεις για τους χόμρεμπόρους σε ό,τι αφορά τα αξιόγραφα. Γιατί? Ξέρουμε ότι μιλάμε για κινδύνους που ξεπερνούν και την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείε οι οποίες και στι ΗΠΑ και στην Κίνα και στην Ιαπωνία δραστηριοποιούνται. Και αν καταργηθούν οι χοντρά αξιογράφων από το πεδίο εφαρμογή τη εταιρεία, τη αυτό θα σημαίνει επιπλέον γραφειοκρατικό άγχο και μάλιστα μεγάλο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι καλά θα κάνουμε να είμαστε επικριτικοί στο σημείο αυτό και θα καταθέσω και σχετικές ε, τροπολογίες και ελπίζουμε να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι ενάφηματα στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστώ. Anybody else? Okay. Θέλει άλλο το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Όχι, ωραία. Λοιπόν, πρώτα πρώτα. Κρίμα που δεν είναι εδώ πέρα ο συγκριτή τη ΕΚΟΝ, γιατί θα έπρεπε να ήταν τέλο πάντων. Οπότε θα έρθει στη συνάντηση των σκιωδών. Αν μπορείτε, δηλαδή ε, σπαθεί μαζί του, να δείτε την εκεί, να τον καλέσουμε τώρα. Έχουμε κάποια βασικά σημεία τα οποία προέκυψαν και σε σχέση με αυτό που είπε ο άντρα και σε σχέση με αυτά που είπε ο, ο και αυτό που είπε ο Πασκάλ πριν. Προσπαθούμε τώρα να πετύχουμε πολλά πράγματα. Μία ένωση κεφάλαια αγορών, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο οι επενδυτές να επενδύσουν και επίσης να είναι πιο εύκολη η προσβασιμότητα των ΜΜΕ στο δανεισμό και στα κεφάλαια. Θυμάμαι και τότε, τότε που ήμουν εισηγήτρια, όλοι λέγανε ότι πάλι καλά που έχουμε αυτή την ρύθμιση, την ευέλιξη να ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να προσφύγουν στην κεφαλαία αλλά τελικά όλη η γραφειοκρατία που είχε ξεκαθαριστεί επανήλθε έτσι είναι ε, αν μιλούμε για έκδοση ομολόγων, χρεογράφων κλπ 5 εκατομμυρίων τότε θα να, να δώσουμε μισό εκατομμύριο για τα έξοδα της ε, γραφειοκρατίας αυτής σε, σε δικηγόρους και λογιστές. Όχι είπα να έχουμε όσο οροφή τα 20 εκατομμύρια για να ισχύσουν αυτά. Ε, και δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί οι περισσότεροι καταναλωτές όταν επενδύουν ε, σε κινητές αξίες Άνοιγουν στη μεσαία κατηγορία, είτε είναι συνταξιδοτικά ταμεία, ό,τι και να είναι. Δεν τα δίνουν χωριστά λίγα-λίγα. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα βαρύ διαδικαστικό οικοδόμημα. Τώρα, η τροπολογία για την έκδοση σε διαφορετικές γλώσσες είχε ζητηθεί από κάποιο φορέα. Έτσι θεωρείται ότι προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές από πλευρά μετάφραση γλώσσα που γράφει το δελτίο. Ανδρέας, ε, κύριε συμφωνείτε σε αυτό που είπατε ότι αφού μιλάμε για retail banking θα πρέπει να είναι ανάλογες και οι ρυθμίσεις να μην είμαστε πάρα πολύ περιοριστικοί, πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά το νοηματικό δελτίο. Αλλιώ πάμε για προσθήκη και άλλη γραφειοκρατία. Η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει, να πει ότι για όλε τι ε, περιπτώσει θα έχουμε πέντε σελίδες παραδείγματο χάρη κλπ. κλπ. Αλλά βέβαια δεν μπορεί, δεν είναι όλοι σε όλε τι περιπτώσει, άρα πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία και την επόμενη φορά που θα ζητήσουμε θα σα πω περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να απλουστεύσουμε την κατάσταση για τι ΜΜΕ. Χωρί χωρίς, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις από την προστασία του καταναλωτού. Ε, ένα καφεδάκι προς το πιούμε πριν έρθει ο Επίτροπος. Καθίστε παρακαλώ. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών. Μιλισμονούμε την προστασία των καταναλωτών. Σκοπός της συναντήσεως να συζητήσουμε την πρόοδο του Προγράμματος Εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις επικείμενες πρωτοβουλίες. Ανταλλαγή απόψεων επί της προόδου. Έχουν ήδη παρουσιαστεί κάποια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες δεν έχουν εγκριθεί ακόμα. Θέλουμε να κατανοήσουμε ποιες άλλες προτεραιότητες θα έχετε στο... και τον υπόλοιπο χρόνο και του χρόνου. Ο Επίτροπος έχει στη διάθεσή του μία ώρα. Και θα σας δώσω λοιπόν το λόγο να κάνετε την παρουσία σας και μετά γίνεται αλλαγή απόψε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Φόρτ, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να σας μιλήσω. Θα σας δώσω, θα κάνω μια αναδρομή πάρα πολύ σύντομη και μετά θα αναφερθώ σε μελλοντικές ενδεχόμενες συζητήσεις για το επόμενο εννιάμινο, δωδεκάμινο. Λοιπόν, έχουμε τη συμφωνία που επετεύχθη για την ασφάλεια των πληροφοριών και το δίκτυο, την ε, οδηγία NICE και βασιστήκαμε σε αυτήν για να δημιουργήσουμε την πλατφόρμα ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, για την κυβερνοασφάλεια και πώς εντάσσεται στον ορίζοντα 2020 και σε συνάρτηση με τις άλλες σχετικές δραστηριότητες, δηλαδή θέλαμε να πετύχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, ασφαλής των δεδομένων. Γνωρίζετε το πακέτο TSM και συμπεριλαμβανόμαστε λοιπόν. Είμαστε στη φάση λοιπόν της πρόσβασης χωρίς ε, φραγμούς, όπου την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα τρομερή διάλογο για τις δυνατότητε ε, του Συμβουλίου να πετύχουμε με τη δική μας υποστήριξη μια επιτυχία στον κλάδο αυτό. Χθέστε στην Επιτροπή. Κοιτάξαμε το πακέτο το, της, ε, του Digital Industry. Το θέμα λοιπόν τι είναι. Πριν από ένα χρόνο στο Ανώπερο, στην έκθεση, κάναμε μία διάλογο με τη βιομηχανία και με τα συνδικάτα, με τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τα, την αξιοποίηση των εφιστάμενων αυτών εθνικών δικτύων, ε, όπως στη Γαλλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Γερμανία. Και θέλουμε στον δρόμο της ψηφιοποίησης ε, της πραγματικής μας οικονομίας να θίξουμε τα θέματα τα οποία έχουν πραγματικά προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Θέλουμε με το πακέτο αυτό τα εθνικά αυτά δίκτυα να τα αναπτύξουμε. Θέλουμε να κοιτάξουμε μια σειρά, ένα κατάλογο τυποποίησεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις υπηρεσίες τυποποίησης και θέλουμε να κοιτάξουμε τα βήματα τυποποίησης και να τα επιταχύνουμε για τον κλάδο αυτό. Προσπαθήσαμε να, κοιτάξουμε το θέμα της συνδεσιμότητας και της δυνατότητας και ανάγκης μετάφορας ε, σε ό,τι αφορά την μετάβαση προς την κοινωνία του Gigabyte. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε και να συγχρηματοδοτήσουμε μάλιστα μια ευρωπαϊκή υπηρεσία προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο τα επόμενα χρόνια και να δώσουμε πρόσβαση σε όλους τους ερευνητές, τους επιστήμονες που υπάρχουν. Έχουμε ευρωπαϊκά κονδύλια. για επενδύσεις ε, high performance computing ε, με απότερο σκόπο να <coughs> συγκεντρώσουμε τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουμε επίση ομίλους από διάφορα κράτη-μέλη και από διάφορες έντρες, ε, για παράδειγμα στη Στουτγκάρδη, τους οποίους, ε, με τους οποίους συνομιλούμε προκειμένου τα επόμενα δύο-τρία χρόνια να μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσεις ε, σε τέτοιες προς κατευθύνσει. Αυτό το χθεσινό λοιπόν πακέτο θα παρουσιαστεί σε μια διάσκεψη στο Ανόβαρο και θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση του δομημένου διάλογου με την κοινωνία, με τα συνδικάτα, με τους επιστημονικούς κύκλους, προκειμένου όλα αυτά τα έργα ε, να προχωρήσουν προς την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας μας. Το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαβουλευτεί για ένα πακέτο ηλεκτρονικού εμπορίου και θα αποφασίσει σχετικά. αποκλεισμός, Υπηρεσίες ε, παράδοσης ταχυδρομικών πακέτων και κατά πόσον υπάρχει ανάγκη ρύθμιση στον κλάδο αυτό οπτικοακουστικές υπηρεσίες και σχετικές οδηγίες, η οδηγία για την τηλεόραση, για παράδειγμα, στον ψηφιακό κόσμο και θα αποτελέσει μια πρώτη ανακοίνωση που θα βασιστεί στις διαβουλεύσεις για το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη α, ρύθμισης για την πλατφόρμα α, την επιγραμμική. Γεωαποκλεισμός. Θεωρούμε ότι στον εμπορικό κλάδο στο e-commerce, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, υπάρχει ανάγκη ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί ο καταγερματισμό των αγορών και να υπάρχουν τεχνικές και νομικές βάσεις προκειμένου όπως μπορεί κανείς να μπει σε ένα μαγαζί στο Μπορντό ενώ είναι από την Βαρσοβία να μπορεί να το κάνει το ίδιο και online. να μην ε, τον παραπέμπουν στη Βρέμη για παράδειγμα ή κάπου αλλού. Θέλουμε οι έμποροι της Ευρώπης να μην υποχρεώνονται, μην υποχρεούνται να ε, ενεργοποιούνται και να λειτουργούν ευρωπαϊκά. Αλλά θέλουμε στο διαδικτύο οι τεχνική φραγμοί που υπάρχουν τώρα και δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο να μην διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. Η οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Από το 2007 που εγκρίθηκε έχουν αλλάξει πάρα πολλά σημεία σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και εδώ οι κλασικές, ε, τα κλασικά κανάλια, το BBC, ARD, ZDF, RTL και ούτω καθεξής. Η γνωστή παροχή streaming, Spotify, Amazon, YouTube και νέους ε, φορείς. Έχουμε την προστασία της νεολαίας εδώ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως αξία, η περιορισμός και η πάταξη των ε, ομιλιών μίσους, ε, το θέμα της διαφήμισης να το κοιτάξουμε και το κατά πόσον ε, αυτές οι υποχρεώσεις μπορούν να συνεχίσουν να παραμείνουν χωρίς ειδική ρύθμιση. Χρειαζόμαστε κανόνες επίσης για την εύκολη πρόσβαση του καταναλωτή σε κάποιες ε, τηλεοπτικές υπηρεσίες. Ναι ή όχι. Βρισκόμαστε σε φάση λοιπόν αναθεώρησης και χρονισμού της οδηγίας. Τις επόμενες 8 εβδομάδες ε, θα καταθέσουμε νομοθετική πρόταση. Στο θέμα λοιπόν αυτό έχω ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να παρουσιάσω επειδή αλλάζει πολύ γρήγορα ε, το οπτικοακουστικό πλαίσιο, αν ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία πρόταση σε ένα-δύο χρόνια και χρειαζόμαστε τρία χρόνια μέχρι να περάσει από διαβουλεύσεις και να εφαρμοστεί τελικά στα εθνικά κράτη-μέλη η νομοθεσία και θα έχει αλλάξει ο κόσμος το 2019. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα αυτό σε βάθος αλλά και πάρα πολύ γρήγορα. Την Σλοβακία και τη Μάλτα, τους επόμενους δύο προέδρους του Συμβουλίου, τους έχω ζητήσει να διαβουλευτούν για το θέμα αυτό, γιατί ο ψηφιακό κλάτος χρειάζεται δις, ε, γρήγορες αποφάσεις για την ε, ρύθμιση ή τα άλλως άμα οι διαβουλεύσεις τραβήξουν σε μάκρο, τι νόημα έχει η τ αμα οι διαβουλευσεις τραβηξουν σε μακρο τι νοημα εχει η ρυθμιση οι δημόσιε διαβουλεύσει για το θέμα των πλατφόρμων online θα... που ολοκληρώθηκε μάλλον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά μέχρι τέλη Απριλίου γιατί είναι πάρα από χίλιε συνεισφορέ. και μέχρι μέσα Μαΐου θα έχουμε δημοσιεύσει, θα δημοσιεύσουμε τη σχετική αξιολόγηση. Και υπάρχει μια βαθμία προσέγγιση από πλευρά μα. Εκεί που έχουμε λέξει specialis, ή θα αναπτυχθεί λέξεις σπεσιάλες όπως για παράδειγμα στο αναθεώρηση του Telecom, στο copyright. Θα προτείνω ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά και το τρίτο τρίμηνο του έτους θα κληθούμε να αποφασίσουμε κατά πόσον και πέρα από αυτό υπάρχει γενική ανάγκη ρύθμισης ή κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι όχι, πέραν από αυτά θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες των, ε, της πλατφόρμας online θα συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου, της απαγόρευσης ε, διακριτικής μεταχείρισης και ούτω καθεξής. Το ερώτημα του κατά πόσο υπάρχει ανάγκη γενικής αντιμετώπισης και γενικής ρύθμισης θα το κοιτάξουμε το φθινόπωρο αξιολογώντας τα υπέρ και τα κατά. Και σε ό,τι την αναθεώρηση του πακέτου TSM, βρισκόμαστε στη φάση αναθεώρηση του πακέτου TSM σε ό,τι αφορά το πακέτο για το roaming, για τους χονδρεμπόρους και τον Ιούνιο του 2016 θα υποβάλουμε μία πρόταση προκειμένου τον Μάιο του 2017 όταν θα καταργηθεί τελείω η περιεγωγή να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτά που επιθυμούμε για την κυβέρνηση ασφαλεία. Το ανέφερα αυτό εν συντομία. Οι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά θα πρέπει να σκοπό έχουν την ενίσχυση της ασφάλειας ε, του κυβερνοχώρου και έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και μέσα από τον ορίζοντα 2020 σε ό,τι αφορά τα νέα έργα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και για μας τους επόμενους μήνες είναι ο έλεγχος του πλαισίου τηλεπικοινωνιών, αναθεώρηση του τομέα τελκο τηλεπικοινωνιών. Θέλουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το φθινόπυρο, να υποβάλουμε μία πρόταση αναθεώρηση, εξυγχρονισμού. Και ποιο θα είναι το θέμα. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όποιος περίπου πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε την απελευθέρωσή του, και ο οποίο ζει από τον ανταγωνισμό, όχι από την μονοπόλια. Το θέμα λοιπόν είναι καταρχά να δούμε πώς μέσω της να νομοθεσία μπορούμε πιο πολύ από ό,τι έω τώρα να δώσουμε κίνητρα για τι επενδύσεις στις ψηφιακέ ε, υποδομές ε, στο βριζονικό φάστα. Θα πρέπει να γίνει μια τέτοια επέκταση στην Ευρώπη και αυτό είναι σε ύψος, σε ύψη τέτοια που δεν πρόκειται να τα πετύχουμε με τα κονδύλια ή με το σχέδιο Juncker κτλ. 80-90% θα πρέπει να έλθει από την ίδια την αγορά, από τον ιδιωτικό κλάδο, από τις εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Άλλο θέμα. Το θέμα για την πολιτική για το φάσμα. Στον δρόμο προς την πέμπτη γενιά, στα δίκτυα, κινητά δίκτυα πέμπτης γενιάς. 5G. Χρειαζόμαστε κάποια μέτρα. Καταρχάς, έρευνα. Να συνεχιστεί η έρευνα και να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό συνδέεται και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε ό,τι αφορά το 5GPP. Κατά δεύτερον, συμφωνίε ε, να συναυτούν με άλλε αγορέ όπω αυτή τη Ιαπωνία, τη Κίνα, τη ε, Νότια Κορέα. Έχουμε μια κοινή διακήρυξη και Είμαστε σε φάση διαπραγμάτευση με την ΙΠΑ τη Βραζιλία κτλ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλε μάρκε οι οποίε λοιπόν θα θέσουν τα πρότυπα για τις επόμενα χρόνια. Δεν ε, μπορούμε πραγματικά παρά να τονίσουμε ξανά και ξανά τη σημασία του 5G στο σχετικό συνέδριο στην Παρσελώνα, στη Βαρκελόνη Ουσιαστικά δύο θέματα ήταν αυτά που κυριαρχήσαν, η ασφάλεια και το 5G. Όλες αυτές οι νέες υπηρεσίες, ε, ή e-health, ε, connected trucks, connected cars, αυτοματοποιημένη οδήγηση, όλα αυτά χωρίς ε, μεταφορά πιο πολλών δεδομένων δεν θα είναι δυνατά. Ούτε το 3G, ούτε το 4G το πετυχαίνει, αλλά ο συνδυασμό 5G, 4G και LTD θα μπορέσει να δώσει την απαραίτητη υποδομή. Για την εκχώρηση των συχνοτήτων 5G χρειάζεται κατεπηγόντως δε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσο οι εθνικές αρχές ε, οι δημόσιες αρχές από μόνες τους, χωρίς συντονισμό, κάνουν αυτές τις ε, αναθέσεις σε ό,τι αφορά τις συχνότητες. Δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε συντονισμένο 5G και δεν θα ξεπεράσουμε τις εθνικές τα εθνικά προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμό της πολιτικής για το φάσμα σε ό,τι αφορά το, την αθεώρηση των τηλεπικοινωνιών. Έχουμε λοιπόν μια σειρά μέτρων τα οποία και προβλέπονται για τις ρυθμιστικές αρχές. Είναι απόλυτα σαφές ότι τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό δρόμο Παρά το γεγονό ότι σε ένα ψηφιακό κόσμο θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά στον ενεργειακό κλάδο, για παράδειγμα, ε, στον τραπεζικό κλάδο, στις ασφάλειες, στις γενικές οικονομικές υπηρεσίες, οι ρυθμιστικές αρχές συντονίζονται πολύ πιο πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον ενεργειακό κλάδο, για παράδειγμα, η ΆΖΟ έχει πολύ πιο πολλέ αρμοδιότητε από ό,τι αντίστοιχη υπηρεσία σε ό,τι αφορά τι civil επικοινωνίε. Άρα θα θέλαμε οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ και οι γενικοί διευθυντέ να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιο πολύ. Και αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο που προκύπτει από τα εθνικά επίπεδα να λάβει το ευρωπαϊκό επίπεδο πιο πολλέ αρμοδιότητε. Και φέτο ε, θα υποβάλουμε μια πρόταση για το e-privacy, για μια οδηγία για το ηλεκτρονικό ιδιωτικό χώρο και πριν το τέλη του έτους θέλουμε να καταθέσουμε μια πρωτα... πρωτοβουλία για την ελεύθερη ροή δεδομένων. Εδώ το θέμα δεν είναι δεδομένα τα οποία καλύπτονται από το βασικό κανονισμό για τα δεδομένα ή από το e-privacy. Μιλάμε για την ελεύθερη ροή δεδομένων, για την οικονομία, για δεδομένα ψηφιακών υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τελευταίο ζήτημα, πάρα πολύ ευαίσθητο. Θέλουμε στο δεύτερο ήμιση. Με το δεύτερο μεγάλο μας πακέτο να υποβάλουμε νομοθετικές προτάσεις για το ψηφιακό πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι τον Δεκέμβριο κάναμε μία μικρή πρόταση σε ό,τι αφορά την δυνατότητα μεταφοράς το portability και τώρα έχουμε το ένα δεύτερο πακέτο. Γίνονται διαβουλεύσεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του εκδότη, για παράδειγμα, όλα αυτά αξιολογούνται. Και το φθινόπωρο θα κάνουμε μία πρόταση εξυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού, αν θέλετε, του πακέτου αυτού των δικαιωμάτων ε, του δημιουργού. Αυτό είναι το πρόγραμμα εργασίας του 2016. <laughs> Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές και μετά τους υπόλοιπους. Ο Ανδρέας Σφαμπ πρώτος. Ευχαριστώ Βίκη, ευχαριστώ Επίτροπε. Τρεις ανησυχίες έχω. Αναφέρθηκαν μέρη στην παρέμβασή σας. Πρώτα απ' όλα, ενσωμάτωση των θεμάτων ασφαλείας δικτύου η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων είναι δύο του δύο νομίσματος. Είναι προφανέ ότι έχοντα ψηφίσει το θέμα την περασμένη εβδομάδα, τον κανονισμό για προστασία των δεδομένων, θα πρέπει η ασφάλεια των δεδομένων να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά και οι συμπράξει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα προτείνεται, θα εξασφαλίσουν να θεσπίσουμε γρήγορα προδιαγραφέ στι ευρωπαϊκές επιχειρήσει, που θα εφαρμοστούν γρήγορα. Αυτέ οι επιχειρήσει λοιπόν που μπαίνουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγία που θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στο Κοινοβούλιο, στι Βρυξέλλε. Αυτέ οι εταιρείε πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ούτω ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσει του Δεύτερον, Μιλήσατε για διάφορες πλατφόρμες. Ε, νομίζω ότι είναι καλή μέρα να μιλάμε για πλατφόρμες, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλι ανακοίνωσε ότι υπάρχει δήλωση ενστάσεων κατά μεγάλη εταιρεία του διαδικτύου σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε πολύ λογικοί, διότι όχι όλε οι διαθέσιμε. Ε, πλατφόρμες είναι μεγάλες, άρα πρέπει να έχουμε μετριοπαθή προσέγγιση στους κανόνες, να εστιαστούμε επί οικονομικής αναπτύξεως, επί καινοτομίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός αυτής. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της θεσινής βιομηχανίας, της παλιάς βιομηχανίας. Είναι πολύ ευρεία πρωτοβουλία για να μην μείνουμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως κάποιες ενώσεις επιχειρήσεων ήδη είπαν ότι το πακέτο του 50 δις για την επόμενη δεκαετία δεν αρκεί. Η ερώτηση τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σας για να σπρώξουμε ακόμα πιο πέρα αυτή την πρόταση. Αυτά και ευχαριστώ. Evelyn Gephardt. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή η οποία πραγματικά περιλαμβάνει πάρα πολλά σημαντικά σημεία όπως και πάντα άλλωστε. Θα ήθελα να θίξω ένα μικρό ζήτημα, το οποίο όμως μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Ένα γερμανικό θέμα ουσιαστικά. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε τι γίνεται. Το θέμα αυτό που αφορά λοιπόν τη Γερμανία και στην τελική ανάλυση θα μπορούσαμε ενδεχομένω έτσι να ανοίξουμε την πόρτη προς την ουδετερο... το, το, ότι δεν θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ουδετερότητα του δικτύου. Βλέπω ότι γνέφεται καταφατικά, καταλαβαίνετε λοιπόν κι εσείς ε, και είναι καλό αυτό. Να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε αυτά που είπε ο κύριος Σφάμπ μόλις. Το γεγονός ότι η ασφάλεια των ροών δεδομένων είναι κάτι το οποίο συνεχώ αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι γίνονται απόπειρες ε, όλο και πιο πολλέ, παραβίαση τη ασφάλεια. Είναι ασφάλεια μεγάλο λοιπόν ζήτημα. σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα δεδομένα των αυτοκινήτων που οδηγούν και αυτό ασφαλώς θα μπορούσε να έχει τη φορά. Ε, αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό ο κλάδο και θα πρέπει σίγουρα να το σκεφτούμε πολύ καλά. Το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω το θέμα του γεωαποκλεισμού. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά με απασχολεί ιδιαίτερο. Και με τα λόγια ενό νέου φοιτητή από τη Στουτγκάρντι θα μιλήσω, ο οποίο πριν από κάποιο καιρό μου είπε. Γιατί κυρία Γκέπχαρτ μιλάτε για διασυνοριακό α, εμπόριο. Εγώ νόμιζα ότι έχουμε νέα αγορά. Είναι λοιπόν σήμερα, δεν θέλουν να ακούνε διασυνοριακό εμπόριο. Θέλουν πραγματικά να λειτουργεί η ιστορική αγορά στον κλάδο αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή η ιστορική αγορά να υπάρχει. Και φυσικά εδώ εμπλέκονται πολλοί οι κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να δημιουργηθούν σε ό,τι αφορά τις πωλήσει και τις συμβάσεις στο διαδίκτυο, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε, όπως είπατε, και πολλές ε, περιττές δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα πραγματικά να αντιμετωπιστούν, όπως η διευθυνσία IP, η πιστοτική κάρτα, η οποία δεν επιτρέπεται σε κάποιες χώρες ε, και πάρα πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ιδιαίτερα για τους νέους που κινούνται και μετακινούνται ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάλτον. Ευχαριστούμε. Τελευταία φορά που τα είπατε με την ECR, κάπως με παρεξηγήσατε. Εγώ θεωρώ παράδειγμα το φάμε ότι είναι ήδη εδώ το μέλλον θα προσοχή να μην το χαλάσετε με προστασία κάποιων συμφερόντων αναλογικό περιεχόμενο ή αποκλεισμό κάποιων υπηρεσιών εγώ ε, μίλησα με τον πρόσωπο τύπου σας και λέει ότι θέλετε να βάλετε κάποιο είδους τέλος σε κάποιες ε, υπηρεσίες ε, ψηφιακές όπως το YouTube. Μα αυτό θα, θα, θα, θα είναι μεγάλο χτύπημα για τα εκατομμύρια που το χρησιμοποιούν. Όποιος καταλαβαίνει το ε, το, το, το, τα ψηφιακά ξέρει ότι είναι εκατοντάδες εκατομμύριων που χρησιμοποιούν το ίντερνετ κάθε μέρα. Δεν είναι καλή ιδέα αυτός ο δασμός. Επίσης ένα άλλο χαράτσι όσον αφορά τις διαδικτυακές πύλες ειδησιογραφίας. Όλα αυτά τα χαρασιά είναι κακά για όλους. Δεν θα έχουν ε, ε, επιλογές οι καταναλωτές, αλλά φύγεται και τους ε, μεγάλους και τους μικρούς της αγοράς των ειδήσεων. Εάν επομένως κάνετε αυτό που σκοπεύετε, θα γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια. Και έτσι δεν θα υπάρχει ποικιλία στις ε, πηγές στο ίντερνετ. Λέτε τώρα ότι θέλετε να καταστήσετε Θέλετε να μην υπάρχουν πια εφαρμογές δωρεάν. Όμως ο κόσμος πάλι κατά εκατομμύρια τις χρησιμοποιεί και τις κατεβάζει. Για πέστε μας, είναι αλήθεια αυτό που ο Γιούγκερ από λίγε μέρες στη, στον αγγλικό τύπο που είπε ότι παραπαρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ζωές του κόσμου. Θα απαγορεύσετε τις ελεύθερες, τις δωρεάν μάλλον εφαρμογές. Θα επιβάλλετε αυτά τα χαράτσια και θα επιβαρύνεται το YouTube και για τον αποκλεισμό. Συμφωνώ γενικά ότι ο κόσμος θα πρέπει να μπορεί διασυνοριακά να αγοράζει. Δεν είναι δυνατόν να αναγκάσουμε τις εταιρείε να πουλήσουν σε χώρες που δεν θέλουν να πουλήσουν. Ε, άμα τις ζωρίσουμε θα κατεβάσουν το ίντερνετ της υπηρεσίας τους αυτής που δεν το θέλουμε αυτό. Τώρα επίση για αυτές τις ιντερνετικέ υπηρεσίε και τα, την, υπηρεσία, την οδηγία για τι υπηρεσίε. Μ' αρέσει το κρίκετ. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σπορ στον κόσμο. όμω και το baseball είναι ένα αξιόλογο σπορ. Και υπάρχει το κανάλι να, άρα μπορείτε να δείτε τα μάτς στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιβάλλεται να υπάρχει ε, ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό περιεχόμενο, δυνάμει της οδηγίας. Να υπάρχει δηλαδή ευρωπαϊκό baseball υποχρεωτικά μου θέλει να πάρει συνδρομή. Αλλά ποιοι θα πληρώσουν για να δουν ευρωπαϊκό μπάσκετμπολ. Οπότε παρακαλώ σκεφτείτε τις συνέπειες των αποφασιών σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και θετικά στο που θέλετε να κάνετε, αλλά μην χαλάσουμε αυτό που ήδη έχουμε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Προχωράμε. Λοιπόν, ελπίζω μέχρι τέλος των θητιών μας να δείξουμε στους πολίτες uh, οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε πολλά σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να εστιαστώ επί δύο που αναφέρθηκαν μόλις πρόσκαιρα, ε, μάλλον επιφανειακά φορητότητα καταρχήν, συμπεριλάβατε στην πρότασή σας μία απέτηση ότι οι πάροχοι θα πρέπει να εξακριβώνουν που βρίσκεται ένας συνδρομητής για να εξασφαλίζουν τα πνευματικά δικαιώματα και πρέπει να είναι λογικές οι απαιτήσει λέτε και να μην οδηγούν σε εντοπισμό ε, και παρακολούθηση του που βρίσκεται ο καταναλωτής. Το καταλαβαίνω αυτό, λένε δύσκολο να συντηρηθεί. Θα μας επιτεθούν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Ποια θα είναι η απάντησή σας εκείνους που θέλουν να αλλάξουν αυτή την ισορροπία. Κυρίως εκείνους που υπερασπίζονται τα πνευματικά δικαιώματα. Για τα συνδεδεμένα οχήματα, τα αυτοκίνητα, συμμερίζομαι την άποψή σας για τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, τα συνδεδεμένα το διαδίκτυο. Ε, για να γίνει η Ευρώπη ηγετική δύναμη σε αυτό, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον τομέα σχετικά με αυτό. Μπορείτε να πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι προβλέπετε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτάσεις θα κάνετε, κατευθυντήρες γραμμές, κανονισμό για τα συνδεδεμένα οχήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσίαση αυτή. Συζητάμε το πρόγραμμα εργασία για το ψηφιακή εσωτερική αγορά και πρέπει να διαπιστώσουμε πάρα πολλέ καθυστερήσει. Καθυστερήσει για το γεωαποκλεισμό. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε η κυρία Γκέπχαρτ. Στην Επιτροπή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το θέμα αυτό στην έκθεση για την ιστορική αγορά. Κάναμε προτάσεις και σε ό,τι αφορά το θέμα των ψηφιακών περιεχομένων και σε ό,τι αφορά και την οδηγία για τους δορυφόρους και για την καλωδιακή. Θα πρέπει να λεφτούν υπόψη αυτά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί είναι και αυτή η οδηγία για την δορυφορική και την καλωδιακή για το φθινόπωρο. Το γεωποκλεισμό είναι ένα θέμα, αλλά ο επίσημος λόγος για την καθυστέρηση ήταν ότι γίνεται διαβούλευση για το θέμα της ελευθερίας ε, και για θέματα τα οποία δεν αφορούν την οδηγία. Το θέμα της συνεργατικής οικονομίας ακούστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξηγήστε μας ότι δεν πρόκειται τι θα γίνει, το sharing economy θα το κοιτάξουμε μόνο στην επικοινωνία για την πλατφόρμα, είναι διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες που δεν αποτελούν όμως τέτοια κοινή οικονομία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, μεταρρύθμιση του δικαίου για τα δικαιώματα του δημιουργού. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια αναβολή. Δεύτερη φορά Έγινε μια πρόταση λοιπόν για, ένα νέο, για μια νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα του δημιουργού και τώρα είμαστε δύο χρόνια αργότερα. Αν το θέμα λοιπόν είναι μόνο οι διαβουλεύσει, οι διαβουλεύσει έχουν γίνει και θα. Ε, αναφερθήκαμε και σε θέματα δεν υπάρχουν νέα επιχειρήματα για την καθυστέρηση αυτή. Είναι υποπτό λοιπόν αυτό, παρά το γεγονό ότι ο πρόεδρο Γιούγκερ είπε ότι το copyright ω τμήμα τη ψηφιακή αγορά θα έχει πρώτη προτεραιότητα. Γιατί περιμένουμε ακόμα λοιπόν, παρά το γεγονό ότι θέλουμε να έχουμε προστασία των δικαιωμάτων, αυτό δεν πρόκειται να το προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Και το πιο σκανδαλώδες ε, θεωρώ στο νέο σχέδιο δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συνθήκη για το Μαρακές σε ό,τι αφορά την δυνατότητα για άτομα ε, με αναπηρία τυφλά να μπορούν να διαβάζουν βιβλία. Αυτό έχει τεθεί σε πάυση, δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Το Δεκέμβριο είχατε πει ότι η πρόταση ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί και ότι καθυστερούσε μόνο και μόνο επειδή θέλετε να το παρουσιάσετε μαζί με την αναθεώρηση του copyright. Τώρα μας λέτε το copyright το Σεπτέμβριο, αλλά δεν θα δούμε τη σύμβαση του Μαράκια. Με πόσο θα περιμένουμε τελικά. Να τελικά θα εγκριθεί αυτή η διεθνή συνθήκη χωρίς συμμετοχή α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομική ένωση όπου υπάρχουν τα πιο πολλά βιβλία σε σύστημα Μπράιχ δεν θα συμμετέχει γιατί κανείς ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο δεν κινούνται. Μα σε τι οφείλεται αυτό και τι πρέπει να γίνει επιτέλους για να επικυρωθεί η συνθήκη του Μαράκης. Ευχαριστώ. Έξι άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Θέλετε να ακούσετε τις ερωτήσεις, να τους ομαδοποιήσετε. Ανά Μαρία Κοράτσα Αυτοί θα είναι οι ομιλητέ. Και Νίκολα. Νίκολα, ναι. Um, λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Ένα λεπτό, λίγο πολύ ο καθένας, για να έχει χρόνο να απαντήσει ο Επίτροπος. Η Άννα Μαρία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε. Εσείς θέλατε πάντα να προωθείτε τον κανονισμό υποστασία των δεδομένων, να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό, να ανοίξουμε το δρόμο για την ψηφιακή αγορά στους καταναλωτές. Δεν έχετε αποχωρητευτεί. Έχουμε επιχειρήσεις που μας λένε ότι προβληματίζονται λόγω γραφειοκρατίας, περιπλοκότητας. Ε, δεν κινούμεθα τόσο να καλυφθούμε για μελλοντικέ εξελίξεις. Έχουμε πάρα πολλές εξαιρέσεις, είναι περίπλοκη νομοθεσία. Όλα αυτά επηρεάζουν ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό μας λένε οι επιχειρηματίες. Επηρεάζει και την ροή δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Είπατε ότι το φθινόπωρο θα παρουσιάσατε κάποιο έγγραφο, πρόταση για την ελεύθερη ροή των δεδομένων. Πρόταση νομοθετικού περιεχομένου θα παρουσιάσετε. Ερώτηση. Κατά κάποιο τρόπο θα βρείτε η κάποια ισορροπία. Στόχος μας ήταν να έχουμε κάτι απλό. Κάτι εναρμονισμένο ένα κανονισμό σωστό που θα πετυχαίνει την ακαιρεότητα που θέλουμε. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Χάσαμε τη φιλικότητα της αγοράς που θα ανοίγει το δρόμο για την ψηφιακή μας ατζέντα. Εξυγχρονισμός ε, των πνευματικών δικαιωμάτων ξεφύγαμε τους ψηφιακούς δίσκους και πάμε στην ε, ροή δεδομένων στο διαδίκτυο, το streaming. Όλοι οι κανονισμοί ακόμα στην Ευρώπη συλλέγουν τέλη, σαν όταν αγοράζαμε CD κάποτε. Ε, David ε, Λοιπόν, αυτό είναι εμπόδιο, όπως είπε και ο David, για την ελεύθερη ροή των υπηρεσιών, ψηφιακών υπηρεσιών. Already. Uh, in very much welcome your, your proposal. Look forward to it. Περιμένουμε την πρότασή σας. Ελπίζουμε να είναι ισορροπημένη, όπως την περιγράψατε, να μην φτάσουμε στα άκρα, να μην πιέζουμε τους πάντες να πουλούν παντού. Έχω πολλά άλλα, με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Και ευχαριστώ ήδη για τις πολλές προτάσεις που έχετε ήδη δρομολογήσει. Ο Ρόμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είπατε στους Πολωνούς να πίνουν Μπορντό από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου που είναι άλλωστε και εκλογική μου περιφέρεια γι' αυτό σας το λέω. Πάντως πέρα από τα αστεία θέλετε, θέλουμε να ψηφιοποιηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, η βιομηχανία η ευρωπαϊκή. Αυτό είναι ένα όραμα πολύ σημαντικό. Θέλουμε αυτό να γίνει για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος, αυτές που ήδη είναι σήμερα εγκαταστημένες στην αγορά, αλλά αυτό είναι πολύ τιτάνιο έργο. Όμως είπατε ότι δεν έχει τους πόρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει ψηφιοποίηση. Κοστίζει. Και ότι θα πρέπει να ποντάρεται σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Όταν υπάρχει, δεν υπάρχει πάντα. Και εκεί θα βάλουν το λιθαράκι του τα κράτη-μέλη. Σας ερωτώ. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποιο ε, είδου ε, δοκιμέ προσωμιώσει, ή αν αυτό είναι ψεύδη πόδο, γιατί έχουμε και το πλάνο, το πρόγραμμα Γιούνκερ. Γιατί τα ακούσαμε, μετά πήγε σκοτάθετρο, ακούμε δύο ε, κουβέντες γι' αυτό. Αυτό το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση ή για άλλη μια φορά το κάθε κράτος μέλος πρόκειται να ασχοληθεί με τα δικά του προγράμματα και θα καλύψει ότι, τα, τα ψηφιακά και όχι μόνο. Οπότε είπαστε μας θα έχουμε επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό θα γίνει μόνο υπέρ κάποιων κρατών και εις βάρος των λοιπόν. Κάνατε προσωμείωση, σχεδιάσατε, μελετήσατε τι θα γίνει, έχετε έρθει σε επαφή για τη σχετική χρηματοδότηση με όλα τα κράτη-μέλη. Πρόεδρος. Thank σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να μιλήσω για τον υγιό αποκλεισμό. Θέλω να μου πει η Επιτροπή πώς θα βρει τη σωστή ισορροπία για να μην καταλήξει σε δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος καταναλωτών να έχουν επιλογές γιατί έχουμε μικρό μήμι ε σε κάποια νησιά που λόγω οικονομικής κλίμακα και μεγέθους δεν μπορούν να μπουν στην ψηφιακή αγορά και να πουλήσουν και στους 28. Μην με παρεξηγάτε. Εγώ είμαι φανδόν υπέρ της ελευθερίας στην ενιαία αγορά. Όμως δεν μπορεί να κάνουμε το ίδιο για όλους. Χρειάζεται διαφοροποίηση. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να καλύψουμε και τους 28. Να μην πετάξουμε ξέρω την αγορά κάποιες ΜΜΕ. Άρα, τι θα κάνετε, πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα το οποίο είναι τόσο δύσκολο, ούτω ώστε να είστε δίκαιοι προς πάντα προμηθευτή και πάντα καταναλωτή. έβα Πολύ χαίρομαι που ήρθατε να μας μιλήσετε κύριε Επίτροπε. Έχω δύο ερωτήσεις. Να, να τις συγκεκριμενοποιήσω όσο γίνεται, διότι είναι δύο σημαντικά θέματα και ευρύτερες σημασίες. Δημοσιοποιήσατε για τον γεωποκλεισμό τις αρχικές σας ε, σκέψεις και συμπεράσματα και ιδίω για τον γεωποκλεισμό στον το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και ήταν εκπληκτικά αυτά που λέτε για τα χαμηλά ποσοστά αγοράς, ε, αγορών τέλο πάντων που γίνονται από την Ανατολική Ευρώπη. Μέσα είναι και η Βουλγαρία η χώρα μου. Και άλλες χώρες εκτός Ανατολικής Ευρώπης όπως το Λουξεμβούργο έχουν νούμερα δέκα φορές πιο μεγάλα διότι εκεί ο κόσμος ασχολείται με διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάμε για 70%. Και εμείς έχουμε 7% στη Βουλγαρία. Και οπότε, μπα και φταίει ο γεωαποκλεισμό για το ότι δεν ψωνίζουν διασυνοριακά ο κόσμος. Άρα, θέλετε να γεφυρώσετε αυτές τις διαφορές με τις νέες προτάσεις για τον γεωαποκλεισμό θα κάνετε κάτι ούτως ώστε να λύσετε το πρόβλημα, ιδίω εκεί που υπάρχει πρόβλημα απλώς πλευρά καταναλωτών με τον διακοσμό. Τώρα κάτι άλλο. Για την ψηφιοποίηση τη βιομηχανία στην Ευρώπη, ε, περίπου ε, αυτά που είπε και ο Ανδρέας Σουβάμπ. Έχουμε πάνω από 30 εθνικές περιφερειακές πρωτοβουλίες για ψηφιοποίηση που ήδη τρέχουν τώρα στην Ευρώπη. Όμως σε κάποιες χώρες όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες για τη βιομηχανία. Άρα, τι θα κάνετε, θα στηρίξετε με κάποιο τρόπο αυτές τις χώρες που δεν έχουν τέτοια προγράμματα και να ψηφιοποιήσουν τη βιομηχανία τους. Για Κονσάρη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ρέντα που είπε ότι η αργή πρόθεση των θεμάτων αυτών μειώνει την αξιοπιστία του σημαντικότητα του προγράμματος που παρουσιάσατε. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά το γεωγραφικό αποκλεισμό. Όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ ταχύες οι εξελίξεις και πολύ δύσκολο βρούμε έναν κανονισμό που να μην δημιουργεί εμπόδια όσον αφορά τις εξελίξεις και την ανάπτυξη. Ταυτοχρόνως όμως, ίσω κάνουμε δραματικά λάθη, τα οποία θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε ίσως, αν προσπαθήσουμε. Ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει έρευνα η οποία μελετά ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Ολιστικά, σφαιρικά, μια πλήρη φωτογραφία. Τι γίνεται στου καταναλωτέ τώρα που ψηφιοποιούνται τα πάντα. Έχουμε ολιστικό όραμα του τι εννοούμε όταν μιλάμε για προστασία καταναλωτών. Okay, Επίτροπε, έχω κάποια σχόλια αν επιτρέπετε. Στους Financial Times σήμερα έχουμε επιστολή 200 Βρετανών επιφανών επιχειρηματιών που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Αλλά θα πρέπει η ενιαία αυτή η αγορά, η ψηφιακή, να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και όχι να την υπονομεύει. Άρα, πώς θα το εξασφαλίσουμε αυτό, πώς θα λειτουργήσουν καλά. Γιατί αναπτύσσει τόσο γρήγορα η ψηφιακή οικονομία. Διότι οι καταναλωτές θέλουν να τη χρησιμοποιούν, τους αρέσει, θέλουν επιλογή, το συνέστημα ότι έχουν ισχύ. Τους αρέσει η ποικιλομορφία που βλέπουν στο διαδικτύο. Όταν μιλάτε λοιπόν για ψηφιακή οικονομία, μπορείτε να μιλήσετε για επιλογή καταναλωτών, ποικιλομορφία, δημιουργικότητα, περιεχόμενο, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό αφήγημα που παρουσιάζεται για τους καταναλωτές που δημιουργούν τις πλατφόρμες, στηρίζουν τις πλατφόρμες, χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Και αν περάσουμε αυτό το αφήγημα, θα θυμηθούμε και γιατί είμαστε εμεί εδώ, σαν Επιτροπή Προστασία Καταναλωτών. Και πρέπει να λειτουργεί η νομοθεσία μα, να το εξασφαλίσουμε αυτό, για την προστασία των δεδομένων. Αυτά που μα έλεγε η Αννα Μαρία, δεν μιλούσε για την νομοθεσία ή την προστασία των δεδομένων. Πρέπει οι επιχειρήσει να έχουν σαφή προσανατολισμό προ να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Να μην έχουμε συγκρούσεις με περχόμενες νομοθεσίες. Όταν εξετάζουμε το θέμα του ψηφιακού περιεχομένου και το δικαίωμα να ζητήσουν οι καταναλωτές για την επιστροφή του περιεχομένου που έχουν ανεβάσει, πώς θα λειτουργήσει αυτό βάσει των πλατφορμών, γιατί καμιά φορά ίσως να υπάρχει κάποια σύγκρουση με την νομοθεσία. Αναφερθήκατε στην ασφάλεια του διαδικτύου, την κυβερνοασφάλεια, αναφερθήκατε σε προδιαγραφές και πρότυπα, το πρωί μια συνάντηση συζητούσαμε στο TTIP, το θέμα του TTIP και φαίνεται ότι καθορισμός προδιαγραφών ε, για την κυβερνοασφάλεια οδηγεί σε διαφορετικές πορείες Ευρώπη και ΗΠΑ. Τι θα γίνει λοιπόν με τις προδιαγραφές. Θέλουμε κάτι καλό ε, όσον αφορά τις κατανοτές και τις επιχειρήσεις, αλλά μην διαφέρουμε. Εμείς χρησιμοποιούμε ISO. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν NEST, NEST, κάτι τέτοιο. Οπότε θα πρέπει να καθοριστούν συμπλέοντες, ε, συμπλέουσες προδιαγραφές. Έχουμε την έκθεση Γκέπχαρτ Κάλλας. Εκεί συζητήσαμε τις διαφορετικές πλατφόρμες, πόσο διαφέρουν η μία από την άλλη. Όταν ομοθετούμε για τις πλατφόρμες όταν κάνετε προτάσεις, σας παρακαλώ, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πλατφόρμες με μεγάλες διαφορές θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν εντός της ποικιλομορφίας οι καταναλωτές και της δημιουργικότητας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε μια δίκαιη ενιαία αγορά η οποία παρέχει την κατάλληλη προστασία στους καταναλωτές. Έχετε 12 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και για τις τοποθετήσεις σας. Καταρχάς, κυρία Ρέντα, δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάτι σκανδαλώδες. Δεν συμφωνώ εγώ δεν ε, προκαλώ σκάνδαλα στο Μαρακές, για παράδειγμα, στην ε, υπηρεσία μου. Αν ε, μου ζητήσει η υπηρεσία μου τρεις μήνες παραπάνω και γι' αυτό λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2016, μετά Χριστό, περιμένουμε το, τη συνθήκη του Μαρακές. δεν είναι σκάνδαλο αυτό, να με συγχωράτε. Θεωρώ ότι η επιλογή των λέξεων ε, είναι καλή για το Twitter, αλλά εγώ ακολουθώ τη συνείδησή μου και την καλή μου πίστη. Έχουμε κάνει περικοπές ε, στις υπηρεσίες μας ε, και είναι μεγάλο το έργο. Κάνουμε ό,τι δουλειά μπορούμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Κάνουμε υπερορίες και για για το συμφέρον των υπαλλήλων μας πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ ότι είναι σκάνδαλο και το Μαρακές, η συνθήκη του Μαρακές θα έρθει το Σεπτέμβριο. Κατά δεύτερον, το σχέδιο εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 θα το ολοκληρώσουμε εγκαίρως. Ε, επιμένω γιατί η πλειονότητα των έργων που περιγράψαμε καταδεικνύει ότι η... σε όλα αυτά τα έργα ενδεχομένω να υπάρχουν κάποιε εβδομάδε, κάποιε μήνε καθυστέρηση, αλλά όλα θα ολοκληρωθούν μέσα στο έτο. Κατά δεύτερον, η χρηματοδότηση όντως 15 ε, δισεκατομμύρια κινητοποιούμε στο πακέτο για την βιομηχανία. Δεν έχουμε πιο πολλά. Δεν μας έδωσε το κοινοβούλιο δηλαδή πιο πολλά. Θα ήθελα να αυξήσω σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις δαπάνες για την έρευνα στη Γεωργία κτλ. Αν σε από τη Γαλλία, θα το κάναμε για το Connecting Europe Facility πολέμησα στου κόλπου τη προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέα δισεκατομμύρια ενέργεια, νέα ε, δισεκατομμύρια για την ψηφιακή. Η Νέλη Κρούς ε, έκανε περικοπέ. Ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το Connecting Europe Facility ένα δισεκατομμύριο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα σε ό,τι αφορά το, την βρυζανικότητα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε παραπάνω λεφτά για τα 15 δισεκατομμύρια. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε θέματα υπόδομων, θέλουμε να συγχρηματοδοτήσουμε τους μεγάλους υπολογιστές σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για το cloud, για την έρευνα, του ψηφιακούς κόμβους, για την αποκεντρωμένη συμβουλευτική προς τις μικρομεσαίες. Θα τα συγχρηματοδοτήσουμε αυτά. Και με τα μέσα αυτά θεωρούμε ότι θα υπάρχει ε, τριπλή συγχρηματοδότηση από εμά, από τα κράτη-μέλη και από την βιομηχανία. Τα κράτη-μέλη και από τα περιφερειακά ταμεία μπορούν ε, να δαπανίσουν ε, πιο πολλά χρήματα για άλλα θέματα από τη στην ψηφιακή οικονομία. Είναι δική τους απόφαση. Δυστυχώς ε, Εμεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να συμμετέχουμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, εκχώρηση των κοντιλίων από τα περιφερειακά ταμεία. Του συστήνουμε κάποια πράγματα, αλλά είναι στην διακριτική του ευχαίρεια το πού θα δαπανίσουν τα ταμεία αυτά. Για την αποδικότητα του ευρυζωνικού φάσματο. κάναμε μια σαφή α, μελέτη και μίλησα για μια κοινωνία γιγαμπάιτ. Η επέκταση προαπαιτεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τι να λέμε για σχέδιο ε, Juncker και για περιφερειακά ταμεία. Σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσον θα δαπανίσουν μεγαλύτερο ποσοστό για την ψηφιακή οικονομία, για την ψηφιακή οδό, πέρα από τις ε, χερσαίες και τις δρομικές οδούς. Και είναι πραγματικά συναρπαστικό το θέμα του vectoring, ε, κυρία Γκέπχαρτ. Λάβαμε τη σχετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γερμανίας. 60 σελίδες. Ως τώρα. Ήμασταν σε συμβουλευτική μορφή. Τώρα έχουμε μέχρι τις 10 Μαΐου χρόνο για να κοιτάξουμε κατά πόσον αυτή η πρόταση ε, απόφαση συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχω οργανώσει μία σειρά κροάσεων τους επόμενους μήνες τις επόμενες εβδομάδες και στις 10 Μαΐου θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει κατά απόψεων θα προχωρήσουμε σε ενδελεχή ε, ανάλυση και μελέτη δύο ή τριών μηνών. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό. Προς το παρόν πρέπει να σας πω ότι κλείνω προς την εξαγωγή αυτής της ενδελεχούς ε, έρευνας για να μην το ξεπετάξουμε το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι τρεις είναι οι βασικοί στόχοι. Κάθε επέκταση του δικτύου είναι καλή, αλλά δεν θα πρέπει να επαναχωρεί και να, κάνει, να υπονομεύει τον, ανταγωνισμό, να μην κινείται προς τη μονοπόληση. Και κατά τρίτον, δεν θα πρέπει να καταστήσει τις ε, επενδύσεις μη ελκυστικές τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα πρέπει να δίνει κίνητρο. Και πραγματικά είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και ακούμε και τις αντιδράσεις όλων των κυβερνήσεων στο Βερολίνο και πραγματικά θα ήθελα να δω πώ θα, προ τα ποια κατευθύνσεις θα κινηθούν. Για την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο, Είπε και ο κύριο Σβάπ ότι ήταν δύσκολο να πείσουμε τα κράτη-μέλη για το ότι θα καταστεί η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα η κυβερνό πολλα Πολλά κράτη-μέλη έλεγαν ότι η ασφάλεια των δεδομένων υπάρχει στην ασφάλεια, στην ιστορική ασφάλεια και να μην σα νοιάζει εσάς Ευρώπη με τα θέματα ε, της νομοθεσίας για τις ροές πληροφοριών έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα και ελπίζουμε σύντομα να κάνουμε αναθεώρηση και να εμβαθύνουμε. Και με το Cyber PPP θεωρώ ότι έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για να πετύχουμε σε ευαίσθητε υποδομέ σε υψηλό επίπεδο ασφάλεια, καταρχά, και κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την βιομηχανία για την ασφάλεια δεδομένων, να την προωθήσουμε προκειμένου να υπάρχει και στον τομέα αυτό μία ευκαιρία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της αγοράς. γεώ αποκλεισμός. Ακούσαμε διαφορετικές τοποθετήσεις εδώ στην αίθουσα. Και αυτό καταδεικνύει ότι ένας έμπορος, ε, για παράδειγμα, κρασιού από την Κύπρο δεν μπορεί να υποχρεωθεί να ικανοποιεί ε, επιθυμίες ε, παραγγελίας από την Ιρλανδία. Γι' αυτό δεν λέμε ότι ο μοναδικό στόχο είναι το άνοιγμα τη αγορά. Απλά δεν θα πρέπει να υπάρχει αδικαιολόγητο γεωαποκλεισμό. Ένα παράδειγμα, αν ένα αγορό κρασιού από τον Πορτό, για παράδειγμα, παραδίδει τα αγαθά του στη Λιθουανία και υπάρχουν ψηλό κόστο, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί. Αλλά γιατί είναι Ολλανδία, δεν είναι αδυνατόν να γίνει άμεση παράδοση, γιατί υπάρχει για παράδειγμα μόνο μία αποθήκη στο Ρότερνταμ. Είναι μεγάλο το κόστος. Αν υπάρχει κάποια δικαιολογία, αν υπάρχει κάποιος λόγος, αν δεν είναι πραγματικά δικαιολόγητος ο γεωποκλεισμός, δεν θέλουμε να βρεθούν σε μειονεκτική θέση οι μικροί. Απλά θέλουμε να είναι ίση η αντιμετώπιση και η μεταχείριση του καταναλωτή. Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παραγγείλει ένα κρασί στο Βέλγιο, αλλά μπορεί να το παραγγείλει στην Ολλανδία. Ενώ ουσιαστικά οι οδοί παράδοση είναι ίδια και δεν υπάρχει άλλο λόγο. Αυτό θέλουμε να αποκλείσουμε για την ελεύθερη ροή δεδομένων. Η επικοινωνία είναι το βασικό ζήτημα στον πυρήνα του ζητήματο σε ό,τι αφορά την κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και με το e-privacy αυτά ρυθμίζονται και είναι θέματα τα οποία είναι οικονομικά και επιστημονικά σημαντικά και υπάρχουν και ρυθμίσεις από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αποτροπή τέτοιας πρόσβασης ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό θέλουμε να αποτρέψουμε. Θεωρούμε ότι η ελεύθερη ροή δεδομένων είναι πραγματικά αναπόσπαστο σημείο της ε, ψηφιακής αγοράς και αυτό θα ε, ενισχυθεί στο μέλλον θέμα της τυποποίησης. Με τη χθεσινή μας ανακοίνωση καταδείξαμε ότι στα ψηφιακά δίκτυα των κρατών μελών σε ποιου τομεί ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει απαραίτητα να γίνει τυποποίηση στα κρατημέλη, στο 5G, στο IoT γενικότερα, στην κυβερνοασφάλεια, Και εδώ θα κινηθούμε και θα συντονίσουμε τη δράση μας προκειμένου να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν ευρωπαϊκά πρότυπα. Βρισκόμαστε σε επαφή με τους Αμερικανούς. Το Σεπτέμβριο μετέβησα στη Washington και ελέγξαμε σχετικούς πίνικες σε ό,τι αφορά το Digital Europe προκειμένου να αναπτυχθούν τέτοια κοινά πρότυπα. Την επόμενη εβδομάδα στο Ανόβρο θα έρθει και η Υπουργό Εμπορίου και για την ψηφιακή, αρχή, ε, ψηφιακή αγορά και θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα τέτοια θέματα για την κοινή αγορά μεταξύ ΙΠΑ και ε, ε, Ευρώπης για την ψηφιακή αγορά. Connected Cars, τα διασυνδεόμενα αυτοκίνητα. Το Σεπτέμβριο του περσινού έτους μίλησαμε με την ΕΣΕΑ και την ΚΕΠΑ τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτέ αυτοκινήτων και με την εκπροσώπους της ε, οικονομίας τηλεπικοινωνιών για να δούμε τι χρειάζεται τα αυτοκίνητα προκειμένου να μπορέσουν μέσω διασυνδεσιμότητας και μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας να λειτουργήσουν τα αυτοκίνητα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι οι υποδομές για την ε, μεταφορά δεδομένων. Δεν έχει νόημα να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, να υπάρχει μια τέτοια λειτουργία, εάν δεν είναι διασυνοριακή ή αν δεν λειτουργεί στην Ήπεθρο. Γι' αυτό το θέμα της ε, συνδεσιμότητας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και των υποδομών για την πραγματοποίηση τέτοιας ε, εφαρμογής των Connected Cars. Τίφεται και το θέμα, για παράδειγμα, της, ε, του δικαιώματος χρήσης των δεδομένων, σε ποιο ανήκουν τα δεδομένα, κατά πόσον όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πακέτο για τα δικαιώματα του δημιουργού θα το παρουσιάσουμε το φθινόπωρο. Στην παρούσα φάση, χωρίς ε, να τσακωνόμαστε για τα αθλητικά και ό,τι θέλετε να βλέπετε. Έχουμε ποδόσφαιρο, baseball, cricket. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Αλλά αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι λαμβάνουμε πολλές αιτήσει για το θέμα, να ελέγξουμε το θέμα των εκδοτών, όχι μόνο των εφημερίδων, αλλά και περιοδικών και επιστημονικών δημοσιευμάτων. και ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν τα πράγματα μεταξύ των εκδοτών, των ε, εταιριών, των καταναλωτών, των δημοσιογράφων. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοια αιτήματα, καλά θα κάνουμε να το ελέγξουμε και έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι σχετικέ διαβουλεύσει, οι οποίε και θα πρέπει να περάσουν από τη φάση τη αξιολόγηση και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα σα διαβιβάσω προτού ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβούμε σε κάποια πρόταση η οποία για σας θα είναι καθοριστική. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να καταστρέψω το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα και να σας πω ότι εγώ δεν υποστηρίζω οποιοδήποτε εκδότη. Είμαι αντικειμενικός, αλλά η, η οικονομική κατάσταση των εκδοτικών οίκων πραγματικά είναι κάτι που με απασχολεί, γιατί δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά. ευρωπαϊκή εκδοτική και η βρετανική όταν μας ε, υποβάλλουν σαφή αιτήματα και αν ε, και οι δημοσιογράφοι, οι ενώσει ε, μα υποβάλλουν τέτοια αιτήματα. Δεν μπορώ να τα πετάω όλα αυτά στο καλάδι των αχρήστων. Θα πρέπει να τα ελέγξω και τα ελέγχω. Και εν γέννη. Στο ψηφιακό ε, χαρτοφυλάκιο. Όταν περνά από την Επιτροπή Κούλ, cool, στην Επιτροπή Ήτρε, από τη Γιούρη, στην ΕΜΚΟ, σε όλο το κοινοβούλιο, σε εσά, σας... Ε, εδώ πέρα με προειδοποιείτε για τους ε, μεν και εκεί με προειδοποιούν για τους δε. Γιατί οι απαιτήσει που μου θέτει η Επιτροπή Πολιτισμού είναι διαφορετική και είναι προ διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι οι δικέ σα ή τη Επιτροπή Βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι σα παρακαλώ Δεν μπορώ να είμαι ε, ο, ο διαμεσολαβητής μεταξύ των επιτροπών και των ομάδων. Θα πρέπει να υπάρχουν συνεκτικές προτάσεις ε, από πλευράς των ομάδων, από πλευράς ε, των επιτροπών. Όσο πιο μεγάλη είναι η συνένεση, τόσο πιο ωφέλιμες είναι οι προτάσεις. Ιδανικά θα ήθελα να υπάρχει μια ψηφιακή επιτροπή, επιτροπή για τα ψηφιακά εδώ στο Κοινοβούλιο. Για να έχω επικοινωνία με μία μόνο επιτροπή και να είναι συνεκτικό ο τρόπο εργασία. Ε, Προ το παρόν είναι αρκετά νομιογενή η κατάσταση εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν το λέω αυτό για να σα ασκήσω κριτική. Η πρόεδρο. Μία διευκρίνηση. Τι είπατε για τι διαβουλεύσει για το copyright και σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες διαβούλευσης, γιατί υπάρχουν ανησυχίε ε, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή. Τι κάνουμε, ε, μήπως έχουμε επιλέξει μόνο κάποιους τομεί για την διαβούλευση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι ξαναξεκινάνε διαβουλεύσεις για το copyright. Και όσοι ήθελαν να καταθέσουν τροπολογίες, ενδεχομένω να μην ακούγονται εξίσου με άλλου φορεί. Πείτε μα με ένα ναι ή ναι, ένα όχι, κατά πόσον έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσει με όλου του εμπλεκομένου φορεί. Κυρία Πρόεδρε, και στην Επιτροπή Μπαρόσο 2, το θέμα του copyright είχε συγκεντρώσει πολλές μελέτες και κάναμε πολλές διαβουλεύσεις, αλλά η Επιτροπή Μπαρόσο 2 δεν κατέληξε σε κάποια πρόταση. Όλες οι μελέτες όμως, όλες αυτές οι διαβουλεύσεις υπάρχουν μπροστά μας, αλλά στην αρχή της δικής μας θητείας είχαμε ανακοινώσει και βάσει των δύο υποθέσεων Google είχαμε πει ότι αναρωτιόμασταν αν υπήρχε ανάγκη ε, ρύθμισης των, ε, της πλατφόρμας ε, online ή κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα πράγματα κατά περίπτωση. Αυτό το ερώτημα τέθησε και σε ακροάσεις, όπου οι παραδοσιακοί φορείς, όπως το BBC, το CDF, RDF, είπαν ότι ε, οι όροι ανταγωνισμού, τι σημαίνουν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι νέοι παράγοντες ανταγωνισμού, οι νέοι φορείς. Γι' αυτό λοιπόν τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο η online πλατφόρμα, ε, για την online πλατφόρμα διοργανώθηκαν διαβουλεύσεις. Και η σκέψη να γίνει κάτι και για τους εκδοτικούς οίκους, μιας και οι ενός εκδοτικών οίκων, πριν από τρεις μήνες ε, μας κατέθεσαν ένα σαφές ερώτημα το οποίο και χρειάστηκε να το αξιολογήσω. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε ε, και εκεί διαβούλευση. Με αυτά τα δύο λοιπόν έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα. Και αυτό θα αποτελέσει τη βάση του προτινόμενου πακέτου. Όλους τους εμπλεκομένους φορείς έχουμε καλέσει να έρθουν σε επαφή μαζί μας για όλα τα θέματα σε όλες τις διαβουλεύσεις Ιούνιο, Ιούλιο, αρχές Σεπτεμβρίου μπορούν να μας υποβάλουν τις συστάσεις τους και να συζητήσουμε εκτενώς αυτές τις συστάσεις για το πακέτο. Σίγουρα θα ακούσετε περισσότερες ερωτήσεις θα θέσουν τα μέλη της Επιτροπής. Όπως ξέρουμε, οι διαβουλεύσεις μπορεί να κλείνει προς μια κατεύθυνση άλλη ανάλογα με την απόχρωση των ερωτήσεων και δυσκολεύουν τα πράγματα αν δεν καλύπτονται όλοι και δεν συμπεραμβάνονται όλοι. Νομίζω ότι είπατε ότι θέλετε να καλύψετε τους πάντες. Θα σας στείλουμε και κάπως διαφορετικά διατυπωμένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ Επίτροπε. Θα προχωρήσουμε, θα συζητήσουμε τη φορητότητα και τη σχετική νομοθεσία. Μάρκο Ζούλο για τη δυσυνοριακή φορητότητα για το υπηρεσίες περιεχομένου διαδικτυακές στην ενία αγορά. Μάρκο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Yes, okay. πρόεδρε. <laughs> Eh, oggi parliamo di portabilità. Μιλάμε για την ε, φορητότητα. Τι θέλουμε να πούμε. Παράδειγμα, αν αγοράσουμε σήμερα DVD στην Ιταλία και το φέρουμε στο Βέλγιο, μπορούν να μου πούν ότι δεν μπορώ να δω το περιεχόμενο. Θα συγκλονιστούμε αν συμβεί αυτό. Διότι έχω αγοράσει κάποια δικαιώματα. Αγόρασα το DVD, αγόρασα τα δικαιώματα και δεν αναγνωρίζω το δικαίωμά μου αυτό. Αυτό συμβαίνει όμως σήμερα. Σχετικά με αυτό, θεωρείται καμιά φορά ότι είναι περιθωριακό πρόβλημα. Τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου όμως μας λένε ότι μόνο το 20% των κοινοτικών ε, ε, επικών έχουν υπογράψει μια σύμβαση για να μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο ε, στο διαδίκτυο. Και μόνο ελάχιστοι από αυτούς περνάνε στο χρόνο στο εξωτερικό πάνω από 10 μέρες. Οι, οι πιο δυναμικοί άνθρωποι της κοινωνίας όμως θέλουν αυτές τις υπηρεσίες εκείνοι που έχουν εκπαιδευτεί στη δυνατότητα ανταλλαγή και στην κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διασυνοριακοί εργαζόμενοι, φοιτητέ που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ένα κομμάτι του πληθυσμού που ε, θα αυξηθεί ε, δημογραφικά. Άρα δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι δεν θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Έχουμε μια δυναμική εδώ όπως είχαμε δει με το roaming, την περιαγωγή. Θεωρούσαμε ότι ένα πρόβλημα αφορούσε λίγους, όμως τα στοιχεία έδειξαν το αντίθετο. Τώρα ξέρουμε ότι χρειάζεται προσαρμογή των ε, κανόνων για μια αγορά που εξελίσσεται τάχιστα. Δεν πρέπει όμως να χαλάσουμε την ευαίσθητη ισορροπία. Δηλαδή, ε, τη, πρέπει να επηρεάσουμε αρνητικά τη χρηματοδότηση του δημιουργού Έχουμε πολύ πλούσια παραγωγή στην Ευρώπη. Οι εθνικές αγορές δεν ε, ταιριάζουν μεταξύ τους. Υπάρχουν γλωσσικές διαφορές, πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Πρέπει να γίνουν σεβαστές. Αν δεν θέλουμε η προσφορά του τελικό χρήστη ε, να ε, μειωθεί. Στόχος είναι η σωστή ισορροπία. Να εγγυηθούμε τα δικαιώματα εκείνων που αγόρασε περιεχόμενο ψηφιακό και ταυτόχρονα να προστατεύεται και η τοπική παραγωγή, να μην πνίγεται η τοπική παραγωγή από τους μεγάλους παραγωγούς. Η φορητότητα δεν θα πρέπει να γίνει σε μια πανευρωπαϊκή άδεια. Πρέπει να γίνει η διακρίση μεταξύ προσβασιμότητας και φορητότητας. Άρα, ποια είναι η συνήθιση διαμονή πρέπει να καθορίσουμε. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Ένα από του στόχου εκθέσεω είναι να εντοπίσουμε ποια από τα κριτήρια μπορούν να μα εξυπηρετήσουν. Να αποφύγουμε καταχρήσει που θα προσφέρει ο κανονισμό και να προβάλλει κανεί εικονική διαμονή. Λοιπόν, χρειάζεται να καθορίσουμε μέγιστο αριθμό ημερών το χρόνο όπου ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φορητότητα. Πρέπει να γίνεται επαλήθευση. Ο πάροχο των υπηρεσιών που πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητα και την πρόσβαση στο περιεχόμενο να μπορεί να γνωρίζει τι γίνεται. Κυρίω τώρα προχωρά γρήγορα η τεχνολογία. Πριν αρκούσε η διεύθυνση του ε, παρόχου IP, τώρα με τα φορητά τηλέφωνα, κινητά δεν αρκεί το IP, η διεύθυνση του διαδικτύου. Λοιπόν, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται σε συνδρομές με πληρωμή, ή δωρεάν συνδρομές όπου προβλέπεται όμως η ταυτοποίηση, η διαπίστωση της ταυτότητας του χρήστη. Πολλές υπηρεσίες σήμερα απαιτούν τα στοιχεία για το χρήστη, αλλά η επαλήθευση δεν γίνεται σε παρκές βάθος. Άρα θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Να προσέξουμε να μην καταπνίξουμε τις ε, υπηρεσίε που παρέχονται στην αγορά. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Πρέπει να τα επισκευαστούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Επανειλημμένα είδαμε ότι το κείμενο δεν έχει στόχο το copyright. Αντιθέτω, αναφέρει στην αρμόνιση των κανόνων τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό εκφράζω τη θλίψη μου και την πικρία μου για την επιλογή να δώσουμε την ηγεσία της εκθέσεως αυτής στην νομική επιτροπή. Είναι μια έκθεση που θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια της Επιτροπής ΙΜΚΟ, διότι είναι σημαντική έκθεση για την προστασία των καταναλωτών. Είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι τα επιχειρήματα που εν γέννη θα συζητηθούν. Με τα χαράς να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους και με τους συζητητές. Στόχος, φιλόδοξο κείμενο, ισορροπημένο, το οποίο να μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι. Η πρόεδρος, από ό,τι γνωρίζω, θα πρέπει να πάει σε μια άλλη συνεδρίαση συντονιστέ του ΙΣΙΑ. Ε, σας πειράζει να αλλάξουμε τη σειρά. Κι εγώ πρέπει να φύγω. Εντάξει. Ωραία, τότε εσείς να μιλήσετε πρώτοι για να πάτε στην άλλη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πρόεδρε και συνάδελφοι. Νομίζω ότι ο κύριος Τζούλο έχει θίξει πολλά από αυτά τα οποία οφείλουμε να ε, συζητήσουμε για αυτή την ε, ε, φορητότητα πολύ σημαντικό για μας της εσωτερικής αγοράς το θέμα γιατί μιλάει για ψηφιακή καινοτομία για το να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο. Γιατί μιλάμε για νόμιμες πλατφόρμες, για νομίμως αγοραστέν υλικό το οποίο έχει κατέλει το διαδίκτυο και έτσι δίνονται κίνητρα στην βιομηχανία να φτιάχνει περισσότερε πλατφόρμες και να εξασφαλίζει ότι ο κόσμος θα έχει την πρόσβαση που θέλει. Ακριβώ όπω είπε και ο εισηγητή, εδώ έχουμε τη λεπτή ισορροπία που πρέπει να εξασφαλίσουμε γιατί είναι ιδιαίτερο ε, σημαντικό όσον αφορά τον ενάρετο θετικό κύκλο. Κίνητρα με τη σειρά τους δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο. Να μην έχουμε έναν στενό κορσέ ε, καταπιστικό και να βοηθήσουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία συνάδουν και έτσι να υπάρχει και η πρόσβαση στο ποιοτικό περιεχόμενο το οποίο είναι και νομίμως αγοραστέν. Άρα, να μην είμαστε πάρα πολύ περιοριστικοί, θα πρέπει να έχουμε νομική σαφήνεια και επίσης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή και στο θέμα του τόπου διαμονής και θα πρέπει με αυστηρό τρόπο να μπορούμε να επαληθεύσουμε, να ελέγξουμε τι γίνεται όσον αφορά τον τόπο διαμονής και κατοικίας. Πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό, διότι α, είδατε τι γίνεται με το νούμερο που πολλές φορές ο κεντρικό κώδικας δεν αρκεί. Γιατί 6.000 ε, είναι αυτοί που λένε ότι μένουν στον Buckingham Palace. Άρα θα πρέπει με αυστηρό τρόπο να γίνεται η επαλήθευση. Και να δούμε με ποιο τρόπο που να είναι και ευέλικτος αυτός τρόπος να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει από χώρα σε χώρα με την κατάλληλη μέθοδο. Αλλά πάντως θα και να αναλογιστούμε τι γίνεται και με την περίοδο εφαρμογή εξάμηνο, δεκαοχτάμηνο, δύο χρόνια. Οπότε μαζί να κάτσουμε να το σκεφτούμε και έτσι να προκύψει μια στεγανή έκθεση της Επιτροπής μας που να αντικαθρεφτίζει αυτό που θέλουμε. Και έτσι σε νόμιμο περιεχόμενο να έχουν πρόσβαση οι ε, επιθυμούντες αυτό καταναλωτές. Η σωστή ισορροπία. Άρα περί αυτού θα τα βρούμε με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε Εύα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ την ε, Επιτροπή γιατί είναι πάρα πολύ προσεκτικά διευκολυνμένο το κείμενο και πάλι και εγώ το βλέπω πάρα πολύ θετικό το να έχουμε μετά την οδηγία έναν κανονισμό πάρα πολύ σημαντικό και οι προτάσεις ε, ακριβώ στοχεύουν σε αυτήν την φορητότητα και αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη όλοι οι συνάδελφοι όταν κατεβάσουν κάποιε τροπολογίε. Πρόκειται για ένα κείμενο σχετικά σύντομο. Πρόκειται για κάποιε προκλήσει τεχνολογικέ ε, και νομίζω ότι το καθήκον μας εδώ ω βουλευτέ και ω μέλη τη επιτροπή είναι να καλύψουμε τι ανάγκε των πολιτών και των επιχειρήσεων. Περί αυτού πρόκειται για αυτόν τον κανονισμό. Να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από τους πολίτες. Αυτό που έχουν αγοράσει νόμιμα. Όταν ταξιδεύουν και ταυτόχρονα οι επιχειρήσει να μπορούν να διευρύνουν το βεληνικέ των υπηρεσιών που παρέχουν χωρίς επιπλέον κόστος η γραφειοκρατία. Να καινοτομήσουν οι επιχειρήσει, να προσθέσουν και άλλε υπηρεσίε προ του χρήστε και οι startups και οι μικροεταιρείες και οι ΜΜΕ εδώ καλύπτονται. Και όλα αυτά να μου γίνει πραγματικότητα μέχρι το 2017. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε μια πρωτοπόρα στοχευμένη δράση χωρίς να απονευρώσουμε την ε, πρόταση του οικονομισμού. Πέρασε καιρό από που δημοσιεύθηκε η πρόταση κειμένου. Άρα θα πρέπει να πάει συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων επιτροπών. Θα πρέπει βέβαια κάποια σημεία να διευκρινιστούν, αλλά για μένα είναι σημαντικό το να μην χρησιμοποιηθεί η πρόταση για να έχουμε τροποποιήσεις στο δίκαιο του copyright. Θα πρέπει να βρούμε τους σωστού διάβλους, ώστε οι εταιρείε να μπορούν να επαληθεύσουν ε, την κατοικία ή ε, τόπο διαμονή των ε, πελατών του. Είναι καλό να υπάρχει αυτό, αλλά να μην παγώσει η πορεία αυτού του κανονισμού. Λέμε τώρα για τον σύνθητο από κατοικίες. Και αυτό μου φαίνεται κάπως μινιμαλιστικό σαν κριτήριο. Άρα θα πρέπει κάπως να εμπλουτίσουμε το κριτήριο αυτό. Βέβαια με αναλογικότητα και να αποφύγουμε έναν πολύ μακρύ ορισμό. Άρα να έχουμε έναν ορισμό ο οποίος θα εξυπηρετεί τον ε, σκοπό αυτού του οργανισμού. Άρα να δούμε τη διαδικασία της επαλήθευσης. Τώρα όσον αφορά το τι είναι προσωρινό ή την μεταβλητή χρόνο να δούμε πόσες μέρες θα ορίσουμε και, αλλά προσοχή να μην το σχέδιο της διάρκειας τέλος πάντων να μην μας οδηγήσει στο να πάψει να υπάρχει ουσιαστικά η φορητότητα. Πάντως ε, πάλι να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να πετύχουμε και τους τρεις στόχους για τους καταναλωτές, για το roaming, ε, για να δούμε τι γίνεται τον γεωαποκλεισμό, μέχρι το 2017. Επομένως, επίσης, θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να ξεχνάμε ότι ανεβαίνει ο ευρωσκεπτικισμός πρόσφατα είναι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Πώς θα πάρει διασυνοριακά πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις υπηρεσίες και θα συνεχίσουν να συνεργάζομαι αγαστά με, την, ε, με τους άντρους. Κύριε Ντάντη, ευχαριστώ πρόεδρε. Τελικά αρχίζουμε και αυτό το θέμα γιατί εδώ και μήνες. Θέλω να δώσουμε συνέχεια ε, μετά όλη αυτή την κουβέντα για τις αρμοδιότητες δυστυχώς όπως είπε ο κύριος Τζούλο η κυρίως αρμοδιότητα δόθηκε στην νομική επιτροπή. Αλλά και εμεί θα βάλουμε το λιθαράκι μα όσο μπορούμε καλύτερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Και εγώ είμαι πεπισμένο ότι το θέμα αυτό έχει μια σημαντική διάσταση για την ιστορική αγορά και για του καταναλωτέ. Και επομένω θα πρέπει να αναλύσουμε το θέμα. Βλέπουμε εδώ τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε τι πρωτοβουλίες για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα πρέπει να έρθουν οι φραγμοί οι οποίοι συχνά εμποδίζουν τους Ευρωπαίους ώστε να μπορούν ελεύθερα να απολαύσουν εις όλη την αγορά το επιγραμμικό περιεχόμενο νόμιμα και στο χώρο, στην χώρα διαμονής για την Ιταλία έχουμε αυτό το σημαντικό βήμα ώστε όπως θέλαμε να έχουμε ε, την άρση το, του, του, του, γεωαποκλεισμού κάτι που δεν δικαιολογείται στο πρώτο αιώνα. Άρα θα πρέπει να μπορεί κάποιο να απολαύσει τα ενταρνητικά στον τόπο της συνήθω κατοικία και από την άλλη μεριά να καλύψουν του ευρωπαϊκούς σχολούς και περισσότερο ταξιδεύουν και έτσι θα πρέπει να δούμε ότι αυτό είναι μια σημαντική κατάκτηση η νέα αγορά γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένη και στα ψηφιακά μια κατάκτηση επομένω, η οποία αποκτά περισσότερο σημασία μια που πρόκειται να έχουμε και κατάργηση της περιαγωγής σύντομα σήμερα έχουμε πολλούς αλλά πάλι ε, περιορισμένο αριθμό ε, δικαιούχων αλλά βέβαια ε, συνεχίζουν αυτοί να είναι πολλοί και θα έχουν την τάση να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας τονίσω ότι αυτή η πρόταση δεν θα πρέπει να τροποποιήσει το, το, το λεπτό θέμα για τα σχετικά νομοθετήματα για το δικαίωμα του δημιουργού. Και θα πρέπει να δούμε πώς με εύστοχο νομοθέτημα θα καλύψουν αυτά που θέλουμε, δηλαδή τις υπηρεσίες αυτές, νόμιμες κλπ. κλπ. Νομίζω ότι το κοινοβουλευτικό έργο θα είναι πολύ χρήσιμο για να ξεκαθαριστεί, να περιχαρακωθούν κάποια σημαντικά σημεία του σχεδίου οικονομισμού και ο τελικός στόχος είναι το να έχουμε ένα κείμενο σαφές που να εφαρμόζεται εύκολα. Βέβαια, ήταν σωστή η επιλογή κανονισμού και όχι οδηγίε. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα διάφορα σημεία. Θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να συνεργαστούμε γι' αυτά και συγκεκριμένα μιλώ για τον ορισμό τη συνήθους κατοικία, την προσωρινή διαμονή σε κράτο μέλο και τις σχετικές διαδικασίες ε, επαλήθευση. Αλλά και αυτά που λέει το άρθρο 3 που λέει για τους παρόχους υπηρεσιών και τις πληροφορίες σε σχέση με τους καταναλωτές. Θα πρέπει επίσης να δούμε ότι μέχρι το 2017 να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή ταυτόχρονα και με την κατάργηση του roaming. Οπότε να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων, των δικαιωμάτων και των πάροχων. Και ίσως θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες προϋποθέσεις απόλαυση χρήση τέλο πάντων σχετικών υπηρεσιών και θα πρέπει να δούμε πώ θα βρούμε την κατάλληλη λύση για αυτή την πρόταση που αξίζει να υποστηρίξουμε. Um, Morten Lockhart. Morten Lockhart. Um, so who else wants to be? You. Uh, sorry. <laughs> covering for Morton. Is that right? Thank you. Yes. It's a long day. Thank you. Dieter Sharon-Sova for the Liberals. No, it's okay. Uh, thank you. Uh, I think I can be rather brief. Uh, I share a lot of the... Συμφωνώ με τα σχόλια που ακούστηκαν, τα περισσότερα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Σπάνια βλέπουμε κανονισμό με οκτώ άρθρα και οκτώ σελίδες. Αν συγκρίνω με την έγκριση τύπου, έχουμε 90 άρθρα και 400 σελίδες. Νομίζω λοιπόν ότι έκανε πολύ καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνέθλιψε εντός τεσσάρων σελίδων το κείμενο και έχουμε ένα πολύ ορθονομικό κείμενο. Εγώ σαν σκιώδης πρέπει να υπερασπιστώ το κείμενο. Κάποιες τεχνικής φύσης ως τροπολογίες έχω. Μία φορά το άρθρο 3, παράγραφος 3. Ζητούμε τους παρόχους να πούν στο συνδρομητή ποια ποιότητα θα έχει αν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία σε άλλο κάτω μέλος. Μου αρέσει η ιδέα που συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση. Αυτό που αναφέρει στην παράγραφο 2. Ο πάροχος πώς το κάνει αυτό στην πράξη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες ε, εξαρτώνται από τις θέσεις πληροφορίες από πλευράς παρόχου. Δύσκολο να εκτιμηθεί η ποιότητα παροχής εκ των προτέρων, ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Θα θέλαμε κάποια διατύπωση που να λέει όπου είναι δυνατόν ή βάση διαθεσίμων στοιχείων που διαθέτει ο, ο, πάροχος. Στα άρθρο 4 υποστηρίζω την παράγραφο για το νομικό πλαίσιο. Θέλουμε ένα παράγραφο που λέει ότι γιατί δεν εμποδίζεται ο παραχός να δίνει πρόσβαση στο περιεχόμενο που είναι νόμιμο στο κάτω μέλος όπου συνδρομητής προσωρινά διαμένει αν επιθυμεί κάτι τέτοιο η εταιρεία. Άρθρο 5 και τη λογική σκέψεις. Η αδίποτε διατύπωση που αλλάζει την ισορροπία που πετύχαν στην παράγραφο 2 πρέπει να αποφευθεί ταυτόχρονα. Να προσθέσουμε τρεις νέες παραγράφους, είτε εδώ, είτε στο άρθρο 4, είτε στο άρθρο 7 Πρώτα απ' όλα μια παράγραφος που θα λέει ότι ο κανονισμός ή η τροποποίηση της συμβάσεως βάσει του κανονισμού δεν θα πρέπει να δίνει δικαίωμα αποσύρσεως από την σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του κατόχου των δικαιωμάτων και του παρόχου των υπηρεσιών. Ενώ η παράγραφος 1 είναι σαφής ότι οι ρήτρες μη φορητότητας δεν μπορούν να εφαρμοστούν δεν αφαιτεί στη δυνατότητα οι κάτοχοι των δικαιωμάτων απλώς μπορούν να αποσυρθούν από τη σύμβαση με τον πάροχο ή τουλάχιστον το φορητό τμήμα, το φορητό περιεχόμενο που περιέχει τη συμφωνία. Δεύτερον, η παράγραφο, θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Μια παράγραφό που θα λέει ότι αυτέ οι αλλαγέ δεν δίνουν δικαίωμα απόσυρση από τη σύμβαση μεταξύ συνδρομητού και παρόχου. Πιστεύω πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και ο κανονικός επιδιώκει να δώσει περισσότερα δικαιώματα στα άτομα. Αυτές οι αλλαγές όμως δεν θα πρέπει να αποτελούν το κείμενο κατάχρησης από οποιονδήποτε προσπαθεί να ξεφύγει από την σύμβαση για τα τηλεοπτικά. Τέλος, και θέλω συμβολή, συμβουλή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ε, συναδέλφους. Θέλουμε παράγραφο που θα λέει γενικά. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν λόγοι για αλλαγή ή αύξηση των τελών που ζητούν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων για πρόσβαση των παρόχων σε περιεχόμενο ή ε, να παρέχουν ή παροχή περιεχόμενο στους συνδρομητές. Δεν θέλουμε η παροχη περιεχομενο του συνδρομητες δεν θελουμε η φορητοτητα να οδηγεί σε αύξηση των τελών που καταβάλουν οι συνδρομητές Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συνεργασία μου με όλους τους ε, σκιώδεις. Καλώς λέει Πρόεδρος. Φανείς από την ΚΟΕ. Από τους Πράσινους. Τζούλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι το βασικότερο θετικό στοιχείο της έκθεσης αυτής είναι ότι είναι μία αμφιλεγόμενη. Και αυτό το εννοώ ως ε, κομπλιμέντο, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που σχετίζεται με το copyright και νομίζω ότι πιστοποιεί το νομικό έργο της, Ευρωπα... Επιτροπής το γεγονός ότι κατάφεραν να παρουσιάσουν ένα νομοθέτημα το οποίο δεν είναι αμφιλεγόμενο. Και είναι και συνοπτικό και επιλύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για άτομα τα οποία ήδη έχουν προσυπογράψει σε μια υπηρεσία να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν από άλλη χώρα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά τίθεται γενικότερο το θέμα του βιοαποκλεισμού και ότι υπάρχουν άτομα που βρίσκονται γενικά από τη λάθο πλευρά των σύνορων και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στι υπηρεσίε αυτέ και θα υπάρχουν πρόσθετες προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ξεκίνησε ενεργά τη συζήτηση και με τι άλλε επιτροπέ πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να αλλάξουν στην ε, πρόταση αυτή. Κάποιες από τις ευκρινήσεις που ανέφερε και η κυρία Σαράντζοβα, ε, ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολούσε και εμάς είναι το ότι θα θέλαμε να, προσθεθεί μία παράγραφος για το μηχανισμό παρακολούθησης, γιατί αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Η μελέτη αντικτύπου επίση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι η πρόταση θα πρέπει να αναθεωρηθεί μετά από πέντε χρόνια και ίσω αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και στο νομικό κείμενο. Νομίζω ότι συνολικά οι ορισμοί και οι όροι στο κείμενο είναι πάρα πολύ σωστοί. Δεν βλέπω γιατί να υπάρχει χρονικό όριο για την φορητότητα, για παράδειγμα. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε σε αυτό. Μ' ανησυχεί λίγο η πρόταση του Συμβουλίου να εισαχθεί ένα στοιχείο τακτικής επιστροφής στο κράτος μέλος διαμονής ε, στον ορισμό. Αν αναφέρεται λοιπόν αυτή η τακτική επιστροφή στο κράτος μέλος διαμονής, μήπως σημαίνει ότι θα πρέπει να το ελέγχουν αυτό οι πάροχοι των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρόντισε να καταρτήσει την πρόταση με τέτοιο τρόπο που να μην τίθενται ανησυχίε για την προστασία των δεδομένων προκειμένου να υπάρχει διαρκή ανάγκη παρακολούθησης του χρήστη. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν, να μην το αλλάξουμε αυτό, μην αλλάξουμε τον ορισμό του συνήθους τόπου διαμονής με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται έλεγχο των ανθρώπων αυτών από τους παροχούς Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί επίσης κάποια διευκρίνηση για το πώς μπορούν καν οι πάροχοι να ελέγχουν τη χώρα διαμονής. Νομίζω ότι ο πιο ευλογός τρόπος ε, είναι να ελέγχονται οι πληροφορίες οι τραπεζικές. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε και αυτό να υποσκελιστεί και να ανοίγει ο κόσμος ε, λογαριασμού ε, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κοιτάξτε, σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσει ένα VPN σήμερα κανείς από το να ανοίξει 28 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Να είμαστε και λίγο αναλογικοί σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που ενδεχομένω να επιβάλλουμε στους παραγωγούς για πλήρω, για α, υπηρεσίες με επιπληρωμή. Ο έλεγχος τραπεζικού λογαριασμού είναι αρκετός. Και σε περίπτωση ελέγχου του συνήθους τόπου διαμονής με εύλογο και αναλογικό τρόπο. Προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία και ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία προκειμένου να τεθεί σε ισχύ από τον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά υπόθηκαν. Με κάλυψαν. Θέλω να υποστηρίξω την Τζούλια για το τελευταίο που είπε. Είναι πολύ σχετικό αυτό που είπε. Πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να μπορούν να απαιτήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών να ελέγχουν συνεχώς ή να εξακριβώνουν τη φορητότητα ε, του περιεχομένου, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει κατάξη από το συνδρομητή, ελέγχοντας που βρίσκονται. Νομίζω ότι δεν θέλουμε να καταλήξουμε στην κατάσταση κατά την οποία υπάρχει συνεχής ανείχνευση των διευθύνσεων IP από τους παρόχων υπηρεσιών, ούτως ώστε να το ελέγχουν. Ελπίζω λοιπόν να μην είναι αντίθετο αυτό με τους κανόνες για προστασία δεδομένων. Δεν ξέρω για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δουλεύει αυτό, έτσι. Θα πρέπει σίγουρα να το λάβουμε υπόψη σαν μία επιλογή για να αποφύγουμε κατάχρηση της χρήσης των δεδομένων. Okay, Καλώς. Το μόνο που θα ήθελα να πω, Μάρκο, είναι το ίδιο που είπα στην, στον Επίτροπο προηγουμένως. Να θυμόμαστε στο φύγημά μας ότι ένα από αυτά θέλουμε να κάνουμε είναι ότι οι καταναλωτές θα έχουν πράσβαση σε ποικιλία περιεχομένου. Ο κίνδυνο είναι ότι αν είναι λάθο η νομοθεσία, όλοι να μπορούν να πάρουν μαζί του το περιεχόμενο, αλλά να έχουν μικρότερη επιλογή περιεχομένου. Θα πρέπει η επιλογή του καταναλωτού και η ποικιλομορφία και η δημιουργικότητα να προστατεύονται, καθώ και τα πνευματικά δικαιώματα. Να είναι διαθέσιμο και το δημιουργικό περιεχόμενο, ποικιλομορφία περιεχομένου. Είναι εδώ ο Επίτροπο Μάρτιν Πρατ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Α, εδώ είστε. Α, γεια, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και ο Ανδρέας θέλει να μιλήσει, αλλά μιλήστε εσείς πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω και πολλά σε αυτή τη φάση. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής που αντέδρασαν θετικά όσον αφορά το κείμενο. Είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορούμε να σας δώσουμε ενδήποτε βοήθεια. Εξηγήσεις, διευκρινήσεις, συζητήσεις. Να επενθυμίσω κάτι στην Επιτροπή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το θυμίσουμε, ότι είναι θέμα πνευματικών δικαιωμάτων και εσωτερικής αγοράς. Είναι σημαντικότατο να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που θα καλύπτει τους καταναλωτές που πλήρωσαν τη συνδρομή τους και να περνά τα σύνορα χωρίς να το καταλαβαίνουν. Εντοπίστηκαν θέματα, όπως ο συνήθις τόπος διαμονής και εξακρίβωση αυτού. Είναι σημαντικά. Χρειάζεται ισορροπημένη, ευαίσθητη και αναλογική προσέγγιση. Επίσης, συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη περιορισμού της φορητότητας και της προσωρινής χρήσεως της φορητότητας για πολίτες που ταξιδεύουν και που δηλώνουν σαφώς τη χώρα διαμονής. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις ανάγκες φορητότητας των πολιτών της Ευρώπης. Είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής, μπορούμε να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε τρόπο απαιτηθεί. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω και την ε, σκιώδη η συγγήτρια την κυρία Πάνοβα που εξέφρασε με σαφήνεια την άποψη του έλκει το θέμα αυτό και φυσικά διαπιστώνουμε ότι αλλάζει ο κόσμος και φυσικά αλλάζουν και οι υπηρεσίες που παρέχονται online στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων του της και υπάρχουν ε, και κοιτά προς την κυρία Κορατσαμπίλντα κάποιες υπηρεσίες που καταφέρνουν να παρέχουν διασυνοριακά χωρίς πρόβλημα τέτοιες υπηρεσίες και φυσικά υπάρχει και μια σύμβαση μεταξύ της σύμβασης, εκτός από τη σύμβαση μεταξύ του ε, παρόχου και του καταναλωτή υπάρχει και η σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και του παρόχου. Και σε αυτή παρεμβαίνουμε με το νομοθέτημα αυτό. Υπάρχει και η απαγόρευση αναδρομικής ισχύω από νομικής άποψης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε κατά πόσον σε τι συμβάσεις αυτές ε, θα πρέπει να παρέμβουμε και σε τι βαθμό. Αναφέρθηκαν και τα θέματα για το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, ω θέματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, γιατί υπάρχει στη τελική ανάλυση και εθνική ρύθμιση για το αγγλικό υπάρχουν, για το αγγλικό ποδόσφαιρο για παράδειγμα, υπάρχουν ε, Διάφορε ρυθμίσει οι οποίε θα αλλάξουν με το νομοθέτημα αυτό και θα οδηγήσουν σε προσαρμογέ τις οποίες δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε. Θα πρέπει να τι συζητήσουμε γιατί θεωρώ ότι με τον έξω ευρωπαϊσμό της αγοράς σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίες αυτές ε, ε, θα πάψουν να υπάρχουν και εθνικές ε, τέτοιες υπηρεσίες Ιδιαίτερα σε μικρά και μεσαία κράτη-μέλη, όπου δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν να παρέχονται τέτοιε υπηρεσίε και θα υπάρχουν και λιγότερε δυνατότητε χρηματοδότηση. Εγώ δεν είμαι από μικρή χώρα και αναρωτιέμαι σε ό,τι αφορά του άλλου. Αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να το θίξουμε το θέμα αυτό, ότι ενδεχομένω να υπάρχουν τέτοιε συνέπειε. Και σε τελική ανάλυση θα πρέπει να δουν και οι συνάδελφοι τι πιστεύουν για την ε, σε αυτή την οποία και υποστηρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μάρκο, θέλει να πάρει πάλι το λόγο. Θε να επανέλθει. Ναι, ναι, ναι, ναι, συντομότερο. Θα ήθελα απλώ να σα πω ότι ναι, με ενδιαφέρει και εμένα το πώ είναι δυνατόν οι μικροπαραγωγοί να παραμείνουν στην ε, αγορά και όταν ισχύσει ο οργανισμό. Και αυτό επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε μια ανάλυση επιπτώσεων όσον αφορά το κόστος των ε, συνδρομών όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής. Η Πρόεδρος ε, για το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να δουλέψεις ε, βιαστικά. Έχουμε και την προθεσμία της Γιούρη γιατί θα το συζητήσουμε στους συντονιστές. Αλλά κατά πώς φαίνεται η προθεσμία για την γνωμοδότηση θα είναι 25 Μαΐου και 24 ε, Ιουνίου τροπολογίες για να πάει για ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο. Πάντως θα ληφθεί η απόφαση στους συντονιστές. Παρακαλώ όμως βιαστείτε, γιατί ξέρω ότι η νομική επιτροπή βιάζεται. Σας ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε στη συνάντηση των συντονιστών σύντομα γιατί έχουμε υπερβεί το χρονικό όριο.